Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι διερμηνείς, λαμβάνω υπόψη το μήνυμά σας. Και θα σταματήσουμε ακριβώς στις 12.30. Ξεκινάμε λοιπόν τις ε, εργασίες μας και πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση θέλω να καλωσορίσω τους προκυκλημένους του κυρίου Κράμερ, του αγαπητού μας συναδέλφου. Είναι προσκεκλημένοι, είναι ομάδα επισκεπτών από το Υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας. Από τη Βάδη Βιτεμβέργη, από την περιοχή αυτή. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Μεταφορών. Καλώς ήρθατε. Καλή συμμετοχή λοιπόν στις εργασίες μας. Allez, nous commençons. Ξεκινάμε με την ημερήσια διάταξή μας. Λοιπόν, υποχρεώσεις, μάλλον δικαιώματα και υποχρεώσει των ε, επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ο κ. Λιμπάτσκι είχε, είχε αναβληθεί η συζήτηση. Λοιπόν, εγκρίνεται λοιπόν αυτή η αναβολή, αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα να σας πούμε όσον αφορά τις ανακοινώσεις. Ξεκινάμε από το πρώτο σημείο λοιπόν. Δικαιώματα υποχρεώσεις των ταξιδιωτών που χρησιμοποιούν του αναδιατύπωση. Ε, κύριε Λιμπεράτσκι, θα σας δώσω το λόγο. Και μετά οι σκιώδεις ηγητέ. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει το λόγο. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε τον κύριο Λιμπεράσκη. Έχετε το λόγο ως εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. αξιότιμα μέλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Είναι πολύ τεχνικό. Είχαμε πάνω από 630 τροπολογίες που υπευλήθησαν. Είχαμε σχεδιάσει σειρά συναντήσεων με τους σκιώδεις εισηγητές και ακολουθήσαμε το πρόγραμμά μας. Είχαμε αυτές τις συναντήσεις. 20 διαβουλεύσεις έλαβαν χώρα με τους διάφορους ενδιαφερόμενους ε, κύκλους. Υπό διάφορες μορφές έγιναν συζητήσεις, επίσημες, διμερείς, γεύματα εργασίας. Συναντήσαμε και ανθρώπους με αναπηρία. Νομίζω λοιπόν ότι κάναμε όλα όσα έπρεπε να γίνουν δύο από τους ε, σκιώδεις, ο κ. Μουσελίεφ, μέλος του ΕΛΚ και ο κ. Κράμερ, εκπρόσωπος της ομάδας του, ήταν παρόντες σε όλες τις συνεδριάσεις και θέλω να σας ευχαριστήσω αυτούς τους δύο κυρίους. Είναι εδώ και φιλοξενούμενοι του κ. Κρέμερ και μπορώ να σας πω ότι προσεκλήθηκε από έναν εξαίρετο Ευρωβουλευτή που πραγματικά δίνει μάχες για θέματα μεταφορών στο Ευρωκοινοβούλιο. Να σας πω λοιπόν τι συνέβη. Έχουμε κάποιες συμβιβαστικέ που σημαίνει ότι έχουμε αλλάξει ριζικά την περίοδο κοινοποίησεως για ανθρώπους ε, με αναπηρία στις 48 ώρες οι 48 ώρες είχαν προταθεί, αποφασίσαμε να περιοριστεί σε ώρο για μεσαίου μεγέθου σταθμούς και 12 ώρες για άλλους σιδηροδρομικούς ε, σταθμούς. Γιατί? Είναι δύσκολο να σχεδιάσει κανείς ένα ταξίδι 48 ώρες πριν, οπότε αυτό θα σήμαινε έλλειψη προσβασιμότητας ανθρώπους με αναπηρικό καροτσάκι. 12 ώρες, όπως αναφέρεται στην έκθεση, είναι εφικτό για τους σιδηροδρόμους και δεν θα πρέπει να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα οικονομικά ή άλλου είδους προβλήματα. Εδώ συμφωνούμε και με τις συστάσεις της Επιτροπής ΥΜΚΟ μετά από πολλές συζητήσεις επίσης είπαμε ότι δεν θα λαμβάνουμε υπόψη την, ε, τις έκτατες περιστάσεις. Ε, δεν θέλουμε να καταχραστούμε αυτό το σύστημα. Τις περιπτώσεις ανώτερης βίας. Δηλαδή να μην επιστρέφονται τα χρήματα 75% ε, αποζημίωση αν η καθυστέρηση είναι δύο ώρες ή περισσότερες. Ο σκιώδης του ΕΛΚ ζήτησε 100% αποζημίωση για καθυστέρηση δύο ωρών. Έχουμε κάποια διαφορά μεταξύ μας, το παραδέχομαι αυτό για λόγους διαφάνειας. Λοιπόν, μετά όταν χάσει κανείς ανταπόκριση, όταν χαθεί ανταπόκριση, θέλαμε οι επιβάτες να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να ταξιδέψουν με το επόμενο διαθέσιμο τρένο, ανεξάρτητα από την εταιρεία, από το μεταφορέα που προσφέρει την υπηρεσία. Μετά τα αποδήλατα στο τρένο. Εδώ είναι το έτος, έχουμε το έτος πολυτροπικών μεταφορών και αυτή είναι μια αναγκαία λύση και είναι μια λύση που συστήνουμε. Είναι και σημαντικό πολιτικό μήνυμα ε, που πρέπει να στείλουμε. Ε, άλλο σημείο. Μια τυποποιημένη μορφή εγγράφου για διαμαρτυρία ε, επιβατών που ζητούν αποζημίωση, που βάλουν αίτηση αποζημίωση. Θέλουμε συγκεκριμένο έντυπο, τύπο εντύπου ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία είναι τυπωμένο το έντυπο. Είτε είναι 5α είτε 7β να είναι το ίδιο, ανεξάρτητα αν είναι γραμμένο το κείμενο στα λιθουανικά ή τα πορτογαλικά. Το έντυπο πρέπει να έχει την ίδια μορφή. Και πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το εξής πρόβλημα. Ότι το Ευρωκοινοβούλιο ε, θα έχει μια στεναρή στάση. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση ισορροπημένη που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και των μεταφορέων των σιδηροδρόμων και των χρηστών οι χρήστε είναι αυτοί που μα καθοδηγούν και απαιτήσει του. Πράγματι, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και οι συνδρομικέ εταιρείε να μπορούν να παρέχουν την υπηρεσία που συζητούμε. Δεν έχει νόημα να απαιτούμε υπηρεσίε υψηλού επίπεδου αν οι συνδρομικέ εταιρείε δεν μπορούν να τι παράσχουν. Θέλουμε περισσότεροι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τους σιδηρόδρομους όχι μόνο αυτοί που μπορούν να αγοράσουν ακριβές ε, υπηρεσίες πολυτελείας που μπορούν να παράσχουν οι σιδηρομικές εταιρείε. Είπα ότι υπάρχουν κάποιες ε, αποκλήσεις απόψεων, αλλά συναντηθήκαμε με τους κοιόδης και υπάρχουν δύο επιλογές μπροστά μας. Είτε μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία και να εξετάσουμε μια αξιολόγηση αντιχτύπου και μετά να εξετάσουμε και τις επιφυλάξεις που έχουν κάποιοι είτε να βρούμε μια άλλη λύση. Αυτό που με εξέπληξε από πλευρά ΣΕΛΚ ήταν ότι οι διαφορές των απόψεων βασίζεται επί των ευθυνών μεταξύ των τα φορέων των σιδηροδρομικών, εκείνων που παρέχουν την υπηρεσία και εκείνων που ε, είναι ταξιδιωτικά γραφεία ή απλώς πολλούν τα εισιτήρια. Ε, η διαφορά μας όσον αφορά τις απόψεις ποια είναι ότι η ευθύνη θα πρέπει να μοιράζεται μεταξύ του πολιτού του εισιτηρίου και του μεταφορέα. Το ΕΛΚ από την άλλη ασκεί μεγάλες πιέσεις πάνω μας και θέλει ο πολιτής να μην έχει ευθύνη. Οι πολιτές απλώς πολλούν το εισιτήριο για κάποια τρένα και κατά... το κατά κάποιο έχει πολιθεί σωστά το εισιτήριο ή όχι ή αν υπάρχει σωστή ανταπόκριση ή όχι και αν παρέχονται σωστές υπηρεσίες αυτά είναι ευθύνη των σιδηροδρομικών εταιριών. Είμαστε Επιτροπή Μεταφορών και είμαστε υπεύθυνοι για τον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών στο σύνολό του. Αυτά προσπάθησα να σας αναφέρω σήμερα. Δεν ήθελα να σας πάρω περισσότερο χρόνο. Έκανα κάποιες ε, προτάσεις για αλλαγές και τροπολογίες. Προτείνω να αναβληθεί η ψηφοφορία, ούτως ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο να εξομαλύνουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Ανέφερα κάποια από αυτά. Και έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία λύση επωφελή για δισεκατομμύρια επιβάτες εκατοντάδες εκατομμύρια επιβάτες και δισεκατομμύρια που ταξιδεύουν συνολικά. Αυτά και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον κύριο Λιμπεράτσκι. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Κύριε Βαντενκάμπ, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούστε, ο κύριος Λιμπεράτσκι ε, μας έδειξε ότι ότι το ΕΛΚ ε, φαίνεται εδώ κάπως ε, θυμωμένο με βάση τα του Πολυμπεράτσκι και ο κ. Μιζελία που λείπει σήμερα και τον οποίο αντικαθιστώ δεν είναι ικανοποιημένο. Στη τελευταία συνεδρία των σχεδόν εισηγητών που έλαβε χώρα στις 17 του μήνα ε, έδωσε την εντύπωση ότι οι συμβαστικοί, συμβαστικές τροπολογίες είχαν ολοκληρωθεί, ότι υπήρχε δηλαδή συμφωνία μεταξύ του εισηγητή και των σχεδόν εισηγητών. Ο κύριος Μιζελιέ λοιπόν θεωρούσε ότι αύριο θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Όμως, τελικά η ψηφοφορία αναβλήθηκε. Και αυτό βεβαίως ήταν έκπληξη για αυτόν. Θα προτιμούσε σαφώς να είχε λάβει χώρα η ψηφοφορία. Είμαστε κάπως χαμένοι σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες. Υπάρχουν 20, εκ των οποίων οι 8 σύμφωνα με τον κύριο Μιζελιέ τουλάχιστον, δεν αποτελούν αποτέλεσμα των τελευταίων διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια τη διαβούλευση των σχεδόν εισηγητών. Με βάση λοιπόν αυτά που μα είπε ο κ. Λιμπεράτσκι, νομίζω ότι πρέπει να επαναλάβουμε τι είναι αυτό ακριβώ που θέλουμε σε αυτό το φάκελο. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να βάλουμε τέρμα σε όλες τις εξαιρέσεις ε, για το 2020. Θέλουμε να προστατεύονται οι επιβάτες και για τις περιφερειακές υπηρεσίες. Ο κύριος Λιμπεράτσκι μας είπε ότι θέλει να υπάρξει μία αποζημίωση για την καθυστέρηση ε, από 60 λεπτά και πάνω, αλλά εμείς θεωρούμε Ο εισηγητής τώρα μας λέει δύο ώρες μάλλον. Δεν είναι κακή, κακό σημείο κίνηση για τις ε, ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Συμφωνούμε με τον κύριο, Λιμπεράτσκι σε ό,τι αφορά την κατάργηση της ρήτρας ανώτερας βίας ε, και τέλος, σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Λιμπεράτσκι πάντα, ε, για την ευθύνη των πολιτών ε, εισιτηρίων μεταφορικών ε, διαδρομών ε, και την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση από αυτού, πρέπει να το συζητήσω με τον κύριο Μιζολιέ πρώτα. Να υπάρχει ένα σύστημα on-off όταν κάποιος χάνει την ε, ανταπόκρισή του, ναι, να το σκεφτούμε. Αλλά πιστεύω ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς ε, ποιες είναι οι προθεσμίες ε, και ποιες είναι οι διαδικασίες για να μπορέσουν να πάρουν το τρένο. Τέλος, σε ό,τι αφορά για σε ό,τι αφορά τους σταθμούς με πάνω από 10.000 επιβάτες, ε, μιλάμε για τρεις ώρες νωρίτερα, έτσι, εδώ. Και όταν είναι λιγότερο από 2.000, είναι 12 ώρες νωρίτερα που πρέπει να ενημερώσουμε. Ο κύριος Μιζελιέ θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε, ότι μπορούμε να βρούμε μια καλή συμβαστική λύση, όμως επαναλαμβάνω δεν πρέπει εδώ να ενσωματώσουμε πολλά στοιχεία από το Συμβούλιο. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να πει ποια είναι η δική του άποψη και μετά θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στον Τρίλογο. Ο κύριος Λιμπεράτσκι Συγγνώμη, ο κύριος Μιζελιέ θα προτιμούσε να ψηφίζαμε 9 ή 10 Ιουλίου πάντως. Είναι η καλύτερη λύση αυτή. Ευχαριστώ ε, τον κύριο Βαντεκάμ. Παρακαλώ να μιλάτε κάπως λιγότερο διότι έχουμε λίγο χρόνο. Κύριε Ντοστόσκι, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ομάδα της ECR και ο κύριος Παρέμκα, ο κύριος εισηγητής, ε, δεν είναι εδώ σήμερα, θα τον εκπροσωπήσω εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή για την έκθεση και το έργο που έχει επιτελέσει. Όλοι θέλουμε μια ισορροπημένη θέση από πλευράς Κοινοβουλίου. Θέλουμε όμως ε, και η νομοθεσία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επιβατών. Οι νέες αυτές διατάξεις πρέπει να μπορούν να είναι και εφαρμόσιμες για τις εταιρείες μεταφορών και να μην δημιουργούν ένα άχθος ε, δυσβάστακτο. Χρειάζεται λοιπόν μια σαφής ισχυρή διαπραγματευτική εντολή. Η ε, μετάθεση της ψηφοφορίας ήταν μια καλή επιλογή για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τα εναπομείναντα εκρεμή ζητήματα. Το Συμβούλιο δεν ακολουθεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα με εμάς. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, όμως ε, το ECR δεν είναι ικανοποιημένο ακόμα σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσει. Θέλουμε να υπάρχει νομική ασφάλεια και θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια και για τους επενδυτές. Αυτή τη στιγμή οι μεταφορείς μπορούν να χαίρουν κάποιον εξαιρέσεων στο 2020. Δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, νέα ανασφάλεια στους επενδυτές αλλάζοντας τους κανόνες στη μέση του παιχνιδιού. Τώρα για τα κατόφλια και τις αποζημιώσεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και το τι συμβαίνει στον κλάδο στις διάφορες χώρες. Να προσφέρουμε λοιπόν, να υποβάλουμε μια πιο ισορροπημένη πρόταση από αυτού. Υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω προσπάθειας και εργασιών. Ο τομέας των σιδηροδρόμων πρέπει να να, το μεταχειριζόμαστε όπως τους υπόλοιπους τομείς ε, μεταφορών. Τώρα για την ανωτέρα βία, ελπίζουμε ότι στις μελλοντικέ συζητήσεις θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το θέμα της ρήτρα αυτής, καθώς και το θέμα της ευθύνη ε, και για τους πολιτές εισιτηρίων. Η ε, σιδηρόδρομη είναι μέρος τη καθημερινότητάς μας. Ο αντίκτυπος λοιπόν του κανονισμού θα είναι μεγάλος. Θα μας βοηθήσει αυτό να ε, κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά αφού γνωρίζουμε ποιο είναι ο αντίκτυπο. Ο κύριο Ρόντ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι που είναι εδώ η διερμηνείς και θα μπορέσω να μιλήσω και τη γλώσσα μου, τα δανεικά. Είμαι κάπως επικριτικός, ξέρετε, και όταν κάποιος επικρίνει άλλους ανθρώπους, ε, καλό είναι να μένει μετά για να ακούσει τις απαντήσεις. Όμως δυστυχώς πρέπει να πάω στην Επιτροπή Γιούρι μετά. Ε, πάντως, αν φύγω, δεν είναι επειδή με αγενείς ή επειδή θύμωσα, είναι πρέπει να πάω να ψηφίσω στην Επιτροπή Γιούρι, σας το λέω από τώρα. Είναι δύσκολο για μένα να αν να αναγνωρίσω την πραγματικότητα που περιγράφει εδώ ο εισηγητής. Να την κατανοήσω. Αναβλήθηκε η ψηφοφορία. Γιατί? Γιατί υπάρχει τεράστια πολιτική διαφωνία. Και υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ μέρους του εισηγητή να αποδεχθεί την πλειοψηφία, την άποψη της πλειοψηφίας στο μελών. Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια των πραγματεύσεων είδαμε ότι οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι, οι γκουε ε, είναι με την πλευρά των ε, επιβατών και η, ο κ. Λιμπεράσκη και η σύμμαχή του είναι υπέρ των μεταφορέων. Εκεί είναι η διαχωριστική γραμμή και πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί αναβάλλεται η ψηφοφορία. Το πρόβλημα είναι ότι ο εισηγητής δεν θέλησε ε, να λάβει υπόψη του την άποψη της ε, μεγάλης πλειοψηφίας. Είπε ο κ. Βανεκάμπ κάποια πράγματα προηγουμένως. Και δεν, δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου η άποψή μας. Ε, Στι συμβαστικέ προτάσεις. Δεν πρόκειται δηλαδή στην ουσία για συμβαστικέ προτάσεις. Πρέπει να είναι ο κανόνας στα δικαιώματα των επιβατών, όχι η εξαίρεση. Και αυτό ισχύει για όλα τα ζητήματα που συζητούμε εδώ. Είτε μιλάμε για τα άτομα με αναπηρία, είτε μιλάμε για τα εισιτήρια, είτε μιλάμε για τις αποζημιώσεις. Όταν υπάρχει καθυστέρηση πρέπει πάντα να υπάρχει ευθύνη ότι ο επιβάτη θα φτάσει στον προορισμό του. Μου φαίνεται πραγματικά περίεργο που εδώ, σε αυτόν τον οίκο, θέτουμε πολύ αυστηρούς κανόνες που ρυθμίζουν ιδιωτικέ εταιρείε ανά την Ευρώπη. Όταν όμως μιλάμε για κυβερνητικές εταιρείες, για κρατικές εταιρείες, ξαφνικά υπάρχει μια απίστευτη βούληση να τις ικανοποιήσουμε. Πραγματικά θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, διότι γνωρίζουμε, διότι ξέρουμε ότι το Συμβούλιο μετά θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να νερώσει την άποψή μας. Και όπως είπε ο κύριος του ECR, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν αυτές τις κρατικές εταιρείε. Και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτή την επιλογή. Εμείς πρέπει να είμαστε με τους επιβάτες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεκράμερ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και ιδιαίτερα για τα γενικά του λόγια προς εμένα τη στιγμή που έχω και δέκα δικούς μου προσκεκλημένους από, από τη Βάδη Βιντεμβέργη Κάπως ασυνήθιστο αυτό. Να πω λοιπόν ότι όλοι ψηφίσαμε την αναβολή της ψηφοφορίας για να βρεθούν συμβασμοί και κάποιες λύσεις. Και όταν γύρισα στο γραφείο μου, έλαβα διάφορα email από διάφορες ομάδες που μου λέγανε θέλουμε να βάλουμε το τάδε, να βάλουμε το δίνα κτλ. Και όλοι φταίνε γιατί νομίζω δεν πρέπει κανεί να κατηγορήσει του άλλου. Βρήκαμε λοιπόν συμβιβασμό, οπότε ρωτάω γιατί το αμφισβητούμε αυτό τον συμβασμό. Νομίζω ότι η αναβολή ήταν σωστή και θα πρέπει να ψηφίσουμε πάντως τον Ιούλιο, όχι μετά τις ε, διακοπές τις καλοκαιρινές, να αναφερθώ και σε κάποια άλλα ζητήματα, ανωτέρα βία. Να το διαγράψουμε, γιατί αν το κρατήσουμε θα μπορέσουμε ποτέ να το ορίσουμε και θα χρειαστούμε 10.000 δικηγόρους στην Ευρώπη γιατί θα έχουμε πάρα πολλές προσφυγές. Το είδαμε και στην αεροπορία, στην αεροπλογία μάλλον, όπου είχε εφαρμοστεί τέλο πάντων και όταν έχουμε θέμα ανωτέρας βίας ε, είχαμε πολλά προβλήματα, οπότε θα έλεγα να το διαγράψουμε για να βρούμε ένα συμβασμό επειδή είναι σημαντικό να μην υπάρχει αβεβαιότητα, ανασφάλεια και να χάνουν πάντα οι επιβάτες. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούμε να ακολουθήσουμε από άλλους τομείς μεταφορών. Μετά, για τα ποδήλατα στα τρένα. Ξέρετε ότι μου είναι προσφυλές αυτό. Πριν 10 χρόνια ψηφίσαμε μόφωνα εδώ στην Επιτροπή ότι τα τρένα ψηλή ταχύτητα θα έπρεπε να παίρνουν ποδήλατα. Τώρα, οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι που πάνε κατευθείαν στο Υπουργείο στο Βερολίνο λένε ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό μόνο όταν δεν δημιουργεί προβλήματα. Και τελικά δεν έγινε ποτέ και απλά και μόνο αυτό αποτέλεσε ένα πρόσχημα. Τώρα βέβαια βλέπουμε να αυξάνεται ο τουρισμός 20% ετησίως. Έχουμε ευρωπαϊκούς ποδηλατοδρόμους, δίκτυο, αλλά κανείς δεν τους χρησιμοποιεί γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς του ποδηλάτου. Θέλουμε λοιπόν να ισχύει αυτό για τα νέα τρένα, για τα τρένα που θα πρέπει να έχουν επί τούτου ειδικό βαγόνι για τα ποδήλατα και να περιλαμβάνεται και η αντίστοιχη σηματοδότηση υπόθηκε ότι θα έπρεπε να μπορούμε να τα βάλουμε σε όλα τα βαγόνια, αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί με τις ε, αποσκευές και όλα τα υπόλοιπα, τα συμπράγκαλα δεν γίνεται. Οχτώ ποδήλατα πάμε το μέγιστο, ένα τρένο, όχι ένα βαγόνι. Τα υψηλή ταχύτητα τρένα ταξιδεύουν με 60% Οπότε υπάρχει μεγάλος χώρος για τα ποδήλατα. Και στα λεωφορεία αυξήθηκε ο αριθμός των ποδηλάτων από 15 και αναγκάστηκε ο κόσμος, είπα, μάλλον προτιμούσε να πάει από τα τρένα στα λεωφορεία επειδή είχε δυνατότητα να μεταφέρει τα ποδήλατα. Δεν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός, αλλιώς ε, θα χάσουμε επιβάτες. Θέλουμε λοιπόν να ισχύουν οι κανόνες, να υπάρχει αυτό το ενιαίο εισιτήριο και όλο το εισιτήριο ακριβώς θα πρέπει να καλύπτει αυτές τις ευκολύνσεις. Ας πούμε και τα νυχτερινά εισιτήρια θα πρέπει να καλύπτουν αυτή τη δυνατότητα. Και αυτός είναι ο δρόμος, αυτή είναι η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι από το 23 στη σύμβαση για τις αποσκευές και τις μεταφορές θεωρούταν φυσιολογικό αυτό να μεταφερθεί δηλαδή ένα ποδήλατο, να μεταφερθεί ένα ποδήλατο. Σχεδόν 100 χρόνια αργότερα δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε και μου φαίνεται απαράδεκτο αυτό. Τώρα η τομεακή λύση ενδεχομένως θα μπορούσε να αποκλείσει κάποιους φορείς ή κάποιους ενδιαφερόμενους, αλλά αυτό είναι παράλογο. Θέλουμε εδώ να εμπλέκονται όλοι, γιατί νομίζω ότι οι επιβάτες ε, δεν κάνει διαφοροποιήσει. Θέλουν ένα ενιαίο ειστήριο να του πάει παντού στην Ευρώπη. Δεν σκέφτονται με εθνικά στεγανά. Η Κομισιόν έχει κάνει ένα βήμα προόδου στο ενιαίο εισιτήριο. Υπάρχουν όμω κάποια κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν και ίσω θα πρέπει να το κάνουμε αυτό στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών. Εμεί θα θέλαμε να υπάρχουν σε ισχύ ενιαία εισιτήρια γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα, θα ωφεληθούμε πλήρως από τα πλεονεκτήματα του σιδηροδρόμου, περιβαλλοντικά, μεταφορικά και άλλα. Μετά στη Γερμανία να σας πω ότι έχουμε μεγάλη εμπειρία, γιατί 90% περιπτώσεων βρήκαν λύση στη Γερμανία. Και αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, σε αντίστοιχο επίπεδο στην Ευρώπη, πανευρωπαϊκά, αλλά θα ήταν θαυμάσιο. Αν τώρα για τις τρεις ώρες ισχύσει το κριτήριο του σταθμού πάνω από τους 10.000 επιβάτες, θα περιοριστούν κατά πολύ οι σταθμοί αυτοί. Νομίζω στις κατοχώρες ισχύει η καθυστέρηση της μιας ώρας. Οπότε οι συμβασμοί που θα πρέπει να μελετήσουμε στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών θα πρέπει να είναι αξιολογή και να ψηφίσουμε τον Ιούλιο ώστε να ψηφιστεί από την τωρινή θητεία αυτή η οδηγία. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ να περιοριστείτε σαν αφορά το χρόνο μιλίας, κύριε Άντερσεν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, οι σοσιαλιστές κατέθεσαν πολλές τροπολογίες για αυτή την ε, έκθεση. Διαφωνώ με τον κύριο Ρέντερ που πρόκειται να φύγει αν δείτε τις τροπολογίες μας, δεν είναι αλήθεια ότι δεν δώσαμε προτεραιότητα στα δικαιώματα των επιβατών. Διαφωνώ λοιπόν με αυτά που είπε, ιδιαίτερα για την κατανομή ευθύνη μεταξύ μεταφορέων. Και αυτό ισχύει κυρίως για τα ενιαία εισιτήρια και τα πρόστιμα. Όταν αγοράζουν οι επιβάτες εισιτήρια από πάνω από ένα πολιτή. Έστω και αν ο προορισμός δεν είναι ο ίδιος, αυτό πρέπει να προβληματίσει. Και αυτό το λάβαμε υπόψη μας. Οπότε στους συμβασμούς θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι όταν έχουμε ανάκτηση από ένα μεταφορέα σε άλλο πολιτή, θα πρέπει να διευκολύνουμε τη δυνατότητα ανάκτησης του ποσού ή αποζημίωσης. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε και για το νέο εισιτήριο, αν εσείς, ας πούμε, βγάλετε τρία εισιτήρια, κανείς ε, δεν εμποδίζει τους ε, πολιτές να αυξήσουν το αντίτιμο του ενιαίου εισιτηρίου, ακριβώς λόγω αυτού του πολλαπλού χαρακτήρα. Και στην τροπολογία 238 έχουμε παραπομπή στην προστασία που παρέχει η και βελτίωσή τη. Το ίδιο και για το πεδίο. Συμφωνώ με τον κύριο Κράμερ από αυτού ότι θα πρέπει να έχουμε πιο περιορισμένη προσέγγιση για το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Έχουμε πολλέ αποφάσει του δικαστηρίου σε σχέση με τι μεταφορέ ζώων, τι εναέρε μεταφορέ που καταδεικνύονται ότι θα πρέπει να περιορίσουμε το πεδίο. Συμφωνώ λοιπόν με τι προσπάθειες του εισηγητή και θα ήθελα να ζητήσω να το εξετάσουμε αυτό σοβαρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Άντερσεν. Να σας πω. Θεωρώ ότι στην ε, έκθεση αυτή υπάρχει μια διαπίστωση η εξής η Ευρώπη έχει σημειώσει μεγάλη καθυστέρηση στη δυνατότητα για τους ποδηλάτες να μεταφέρουν το ποδηλατό τους στα τρένα. 26% των μετακινήσεων γίνονται με ποδήλατο στις 100 χώρες, 19% στη Δανία, 10% στη Γερμανία. Πώς εξηγείται λοιπόν, συνάδελφοι, σε αυτή την μάζα χρηστών που δεν μπορούν και δεν επιφέρουν συμφόρηση στους ε, δρόμους μας ότι η μεταφορά αυτών των ποδηλάτων θα σταματάει στους ιδρομικούς σταθμούς. Εγώ κατέθεσα η ίδια να υπάρχουν 8 θέσεις ποδηλάτων ανατρένω. Για όλα τα είδη τρένων, μεγάλη ταχύτητα, διοσυναριακά, γαλατάδικα, τα πάντα. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, αυτές τις παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή να κρατηθούν ιδιαίτερες θέσεις για τα ποδήλατα, όπως ακριβώς και να έχουν τα δικαιώματα, όπως ακριβώς και οι κανονικοί ταξιδιώτες, επιβάτες. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και τόσο παράδοξο, ιδιαίτερα να δούμε την εξέλιξη της κινητικότητας, η οποία τίνει προς το ποδήλατο, μάλιστα και στο ηλεκτρικό ποδήλατο. Θα ήταν λοιπόν καλό και ευκταίο να προστατεύσουμε την ποιότητα του αέρα μας, και να προστατεύσουμε και το κλίμα μας. Οπότε σας ζητάω λοιπόν μαζί με την πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών να κάνουμε το σιδηρόδρομο συμβατό με το ποδήλατο και να δημιουργήσουμε θέσεις για τα ποδήλατα στα τρένα. Αυτό είναι καλό για τις μελλοντικές γενιές, οι οποίες θα μας ευχαριστούν σε λίγα χρόνια, αλλά είναι καλό και για τον πλανήτη μας. Να σας πω λοιπόν ότι θα ήταν καλό να στέλνουμε αυτό το μήνυμα από την έκθεσή μας αυτή. Θα συνεχίσουμε τις ε, παρεμβάσεις. Κυρία Κρασφάτερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν τέσσερα σημεία που θα ήθελα να αναφέρω. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι καλό που διαγράψαμε την ρήτρα ανωτέρας βίας. Δεν γίνεται οι επιβάτες να είναι υπεύθυνοι για προβλήματα τα οποία οφείλονται ας πούμε στην κακοκαιρία. Και όπως είπε και ο κύριος ε, Κράμερ, ούτως ή άλλως σε άλλους τομείς μεταφορών οδήγησε σε προβλήματα και σε συγκρούσεις, σε διενέξεις. Μετά, οι αποζημιώσεις για τους περιφερειακούς μεταφορείς. Να πω το εξή ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός περιφερειακή μεταφορία μεταφορέα μεταφορών, αυτό ο ορισμό ποικίλει από χώρα σε χώρα. Οπότε ένα ενιαίο ορισμό εδώ θα ήταν χρήσιμο ώστε να μπορέσουμε να βρούμε συμβιβασμού για κάποια θέματα. Έχω και ένα ερώτημα προ τον εισηγητή. Οι εθνικέ εξαιρέσει σε σχέση με του περιφερειακού μεταφορεί περιορίστηκαν στου 12 μήνε μετά από θέση ισχύ τη νομοθεσία. Γιατί αυτό το 12 μήνο. Μετά, οι εξυπηρέτηση του σταθμούς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό τα δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα να ενισχυθούν και οπωσδήποτε συμφωνώ με την αλλαγή αυτή. Άλλο ένα σημείο που είναι επίσης σημαντικό είναι οι online πολιτές εισιτηρίου να είναι υπεύθυνοι για τα εισιτήρια που πολλούν. Δεν μπορούμε να έχουμε καταστάσεις όπου αυτοί μπορούν να κερδίζουν, να βγάζουν χρήματα, αλλά να μην είναι υπόλογοι για τους κινδύνους που ενέχουν αυτές οι διαδικασίες. Οπότε θα πρέπει να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των επιβατών με μια λογική και ρεαλιστική προσέγγιση. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή και θα στηρίξω τη συμβαστική του τροπολογή. Και θέλετε εσείς το λόγο ξανά. Ορίστε. Πολύ γρήγορα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, λέει και ο Να απαντήσω στον κύριο Κράμερ, που φαίνεται να υπονοεί ότι κάποιοι εδώ δεν υποστηρίζουν ε, τις συμβαστικές λύσεις που βρήκαμε. Πρέπει να πω, όχι, αυτό δεν ισχύει. Αληθεύει ότι το ΕΛΚ και οι φιλελεύθεροι επιστρέφουν για να ξανασυζητήσουν κάποια θέματα ασφαλείας. Θέματα που αφορούν τη μεταφορά των ποδηλάτων. Αυτό διότι οι απόψεις μας δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη στα συμβιβαστικά κείμενα. Δεν είναι ότι δεν στηρίζουμε τις συμβαστικές. Στηρίζουμε κάθε συμβιβασμό, αλλά θέλουμε η θέση μας να αντικατοπτρίζεται στο τελικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κράμερ, λιγότερο από ένα λεπτό για να απαντήσετε διότι εδώ θα διευθετήσουμε τώρα μεταξύ, τη μεταξύ συζήτηση. Κύριε Κράμερ, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα ότι ήσασταν κατά των συμβιβασμών, αλλά είπα ότι είχαμε βρει συμβιβασμό για τη μεταφορά των ποδηλάτων όλοι μαζί. Και μετά από δύο ώρες δύο ομάδες έστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα λέγοντας ότι θέλουν να προσθεθεί κάτι. Όταν συμφωνούμε επί συμβαστικών ε, κειμένων πρέπει να το σεβόμαστε. Το ίδιο ισχύει και για άλλους σε άλλα σημεία. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά το πώς δουλεύουμε. Αν έχουμε κάποια συμβαστική πρέπει να παραμένουμε στα αριά του συμβασμού. Ευχαριστώ κύριος, κύριε Κράμερ. Καλό θα ήταν να πάτε να πει ένα καφεδάκι μαζί, νομίζω. και να βρείτε καλό συμβιβασμό. Ε, λοιπόν, δεν έχετε συγχρονιστεί, αλλά το ίδιο σκέφτεστε. Πού είσαστε, ο κ. Γκρίντελ. Α, εκεί είσαστε. Η κυρία, συγγνώμη, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, λέει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελίζα Πεθκότ Χάουσερ, με λένε. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που διεξάγεται για την πρότασή μας. Κατέδειξε αυτή η συζήτηση ότι τα διάφορα θέματα για τα ποδήλατα και για τις διάφορες ανταποκρίσεις είναι θέματα που συζητούνται και στο Συμβούλιο. Ε, συμφωνούμε ότι χρειάζεται ισορροπημένη προσέγγιση στο τέλος είναι αναδιατύπωση του αρχικού κειμένου. Υπήρχε συμφωνία από τις τρεις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά τα διάφορα τμήματα που θα συζητηθούν όσον αφορά την αδιατύπωση. Θέλαμε στο τέλος να έχουμε απλουστευμένες διαδικασίες για να πετυχαίνουμε γρήγορα αποτελέσματα μέσω της πρότασης αυτής. Ε, συντομία, να αναφερθώ σε αυτά τα εισιτήρια, ε, να το θέμα των ευθυνών. Υπάρχουν πολλά, πολλές λύσεις. Συζητώντας τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν για το θέμα των ευθυνών, αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιληθεί το θέμα των ευθυνών, αλλιώς θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Δύσκολα λοιπόν να μπω σε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Αν χρειάζεται βοήθεια, εξηγήσεις όσον αφορά την πρότασή μας, ε, μην διστάσετε, ζητήστε μας να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Σιγητά, κύριε Λιμπεράτσκι, 1,5 λεπτό έχετε στη διάθεσή σας για να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Κύριε Βαντεν Κάμπ, αγαπητέ μου φίλε. Δεν σχηματίστηκε εντύπωση ότι υιοθετήθηκαν οι τροπολογίες συμβαστικές. Υιοθετήθηκαν. Ε, υπήρχαν, ήταν παρούσες και οι νομικές υπηρεσίες, η νομική υπηρεσία παρούσα και επιβεβαίωσε ότι όλα έγινε σωστά. Με εκπλήσει ότι είπατε ότι δεν ε, δεν είχαμε συμφωνήσει. Είχαμε ανταλλάξει αυτό το θέμα ε, της ανωτέρας βίας και του 70% είπαμε θα αφαιρέσουμε, ε, θα αφαιρέσουμε την ανωτέρα βία για να προστέψουμε την κατάσταση αλλά 75% το συμφωνούμε τελικά. Για την άλλη. Δεν μπορούμε να παραβιάζουμε τις αρχές των μεταφορικών μας συστημάτων. Θέλουμε καλούς σιδηροδρόμους και πρέπει να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο των επιβατών οι σιδηρόδρομοι. Επειδή έχουμε δημόσιους σιδηροδρόμους δεν πρέπει να καταστραφούν και να καταρρεύσουν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε σιδηροδρόμους και πρέπει να λειτουργούν καλά. Δεν αληθεύει ότι ρυθμίζονται ε, σωστά. Πολλές φορές έχουμε υπερβολική ρύθμιση των σιδηροδρόμων. Και αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Μετά. Προτιμώ να συμμετέχουν κάποιοι στις εργασίες και μετά να σχολιάζουν. Ήταν παρόν ο κ. Μουζέλη. Θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η απόψή του. Τόσον αφορά τις εξαιρέσεις. Εγκρίναμε τον εξή συμβιβασμό. Η νέα λύση θα τεθεί σε ισχύ μετά την άρχιση ισχύω του κανονισμού 2022-2024, κάπου εκεί. Αργότερα. Και αυτό λόγω συνεχιζόμενης χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων για τους σιδηροδρόμους όπου αυτό είχε κριθεί αναγκαίο. Χάσαμε την ανωτέρα βία, αλλά θέλαμε να πετύχουμε και μια ισορροπία όσον αφορά τα εισιτήρια πολλαπλών διαδρομών. Αν είναι υπεύθυνη η μεταφορή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για όλα, τότε κάποιοι πολιτές θα πολλούν εισιτήρια με, χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία, θα κερδίζουν χρήματα, αλλά δεν θα είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα της υπηρεσίας που πολλούν. Και δεν θέλω να στηρίξω κάτι τέτοιο. Ο καθένας πρέπει να είναι υπεύθυνο για ένα τμήμα που το αναλογεί της υπηρεσίας. Ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση. Ευχαριστώ για τους επένους που ακούστηκαν. Α, Η Caroline Grand Slider με ρώτησε γιατί χρονική περίοδος για την εξαίρεση είναι αυτή που προβλέφθηκε. Και για τις περιφερειακές μεταφορές αυτό είναι ένα κομμάτι του πεδίου του τετάρτου σιδηροδρομικού πακέτου και των υποχρεώσεων για δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί καθορίζεται τι σημαίνουν τοπικές και περιφερειακές μεταφορές. Αυτά. Έληξε το 1,5 λεπτό μου και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ανεβλήθη για αργότερα η συζήτηση. Προσπαθήστε το μεταξύ να δείξετε συλλογική ε, σύνεση για να βρούμε καλή λύση. Σίγουρα θα καταφέρουμε. Πάμε στο επόμενο σημείο. Επιδοτήσεις για τα καινούργια γιοταχή και διάφορα εμπορικά ελαφρά οχήματα, νέα οχήματα. Η κυρία Κριστίνα Ρεβόλ είναι η συγκήτρια και μετά θα ακολουθήσουν οι σκιώδεις εισηγητές και μετά θα ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Ρεβόνταλόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η γνωμοδότηση έχει 384 τροπολογίες υπευλήθησαν. Έγινε μια συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών στις 5 Ιουνίου. Έχουμε μια νέα συνεδρίαση 26 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί επεξεργαζόμαστε 10 συμβαστικές για τα άθρα 6 ε, ε, και τις αιτιολογικές σκέψεις. Η ψηφοφορία προβλέπεται 10 Ιουλίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος το Σεπτέμβριο από την καθήλη αρμόδια επιτροπή. Πρότεινα συμβιβασμού επί πολλών πτυχών του κειμένου, κυρίως να λάβουμε υπόψη όλες τις εκπομπές και όχι μόνο αυτές από την εξάτμιση και να ενθαρρύνουμε και πιο αντιπροσωπευτικές δοκιμές διότι όλοι θέλουν μια μείωση πραγματική των εκπομπών των ρηπαντικών ουσιών. Όσον αφορά του στόχου του ενδιάμεσου για τη μείωση διοξείδου του άνθρακος το 2025, σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε τύχει συμφωνία, αλλά προχωρούν οι εργασίε. Δηλαδή, το ταχύτερο δυνατόν θέλουμε πριν το 2030 να έχουμε αποτελέσματα, είναι κάτι προ κοινών όφελο η εμπειρία, δηλαδή να βασιζόμαστε μόνο στην καλή βούληση των κατασκευαστών και τη μείωση των εκπομπών όταν δεν είναι νομική υποχρέωση, βλέπουμε στον πραγματικό κόσμο δεν λειτουργεί. Ξεκινώντα από τη διαπίστωση και γνωρίζοντα θα πρέπει όλοι να καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα και καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματο, είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξουμε, συνεννηθούμε όσον αφορά τα μέσα για να πετύχουμε το σκοπό μα. Αντιθέτω, όσον αφορά το επίπεδο των φιλοδοξιών, είναι πιο δύσκολο να πετύχουμε σημείο ισορροπία. Κάτι που να είναι εφικτό και ταυτόχρονα αρκετά φιλόδοξο για να πετύχουμε τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακο προβλέπει η Συμφωνία των Παρισίων αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε ένα αποτέλεσμα φιλόδοξο όσον αφορά τη μείωση του άνθρακο, διότι οι προσπάθειε που δεν θα γίνουν στον τομέα των μεταφορών θα, θα πρέπει να γίνουν αλλού. Όπω στα κτίρια και στη γεωργία. Και εκεί θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και λιγότερο αποτελεσματικά οικονομικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά μεγάλε προσπάθειε από του κατασκευαστέ να προσαρμοστούν στι προδιαγραφέ και να μειωθεί η χρήση άνθρακα από εκπομπή διοξείδιο του άνθρακο από τα νέα οχήματα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μείνουν και ανταγωνιστικέ εταιρείε του παγκόσμιου ανταγωνισμού και να διασωθεί αυτό ο τομέα που επηρεάζει όλη την ευρωπαϊκή οικονομία, όλου τομεί. Θα είναι κάτι σκληρό, αλλά είναι για ε, το καλό τη βιομηχανία και του πλανήτη. Συζήτησα με του κοιόδη ηγητέ. Είναι ένα θέμα περίπλοκο που απαιτεί πολλή συζήτηση. Ε, με με τα χαρά να ακούσω τα επιχειρήματά του όσον αφορά του φιλόδοξου στόχου, του ενδιάμεσου στόχου, όσον αφορά ε, την άποψή του για να μειώσουμε τι κομπές διοξιδίου του άνθρακο από τι μεταφορέ και πώ θα ξεφύγουμε από τη μεγάλη, ε, μεγάλη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτά κυρία Πρόεδρε μέχρι τώρα και επιθυμώ να ακούσω τις απόψεις των διαφόρων συναδέλφων για να βρούμε κάποιες δυνατές συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ κυρία Ραβαντοβολών. Ο κύριος Βιμ Βαντεκάμ έχει το λόγο για το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό το θέμα, ο κύριος Αλήν είναι ο σκιώδης εισηγητής και τον αντικαθιστώ σήμερα και μου έδωσε ένα κείμενο να σας διαβάσω. Και είναι πιο εύκολο έτσι για μένα. Ο κύριο Σελήνη θέλει να ευχαριστήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Πιστεύει ότι αυτό είναι το σωστό επίπεδο για την προσέγγιση που χρειάζεται. Ε, είναι φιλόδοξη στόχη, επιδεικνύει πραγματιστικό πνεύμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρεί και εκείνος, όπως και το ΕΛΚ, ότι είναι σωστέ οι ανησυχίε που εκφράζονται για τι εκπομπέ από τον τομέα των οδικών μεταφορών. Είναι 24% ε, των εκπομπών ε, αυτών των αερίων που προέρχονται από τον τομέα. Και από τα 24% τα 76% των μεταφορών προέρχεται από τι οδικέ μεταφορέ. Ε, πολλά υπόθηκαν για την COP21, για τη Συμφωνία των Παρισίων. Σαν Επιτροπή Μεταφορών πρέπει να συναγάγουμε τα σωστά αποτελέσματα από τη Συμφωνία των Παρισίων και θα πρέπει να κινηθούμε προ μια πολιτική μειώσεω των εκπομπών αυτών, κυρίω στι οδικέ μεταφορέ. Ο κύριο Σαλίνη είναι ανοιχτό, είναι έτοιμο να συνεργαστεί με την εισηγήτρια, ούτω ώστε να καταλήξουν στις σωστές συμβαστικέ λύσεις. Λοιπόν, από πλευρά ΣΕΛΚ θα ήθελα να πω ότι είμαστε κατά της ιδέα της ιδέας να στραφούμε μόνο προς την αυτοκινητοβιομηχανία και να πούμε ότι αυτός ο τομέας είναι ε, αποκλειστικά ε, υπεύθυνο για τη ρήπανση, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Το ΕΛΚ υποστηρίζει την ιδέα μιας προσέγγισης που είναι τεχνολογικά ουδέτερη. Οπότε η μείωση των εκπομπών του διεξιδίου του άνθρακος ε, πρέπει να επιτευχθεί μέσω πολλών μέτρων και πολλών λύσεων που θα πρέπει να εξεταστούν και να εφαρμοστούν. Οι διάφορες τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν θα πρέπει να εφαρμοστούν και πιο γρήγορα και να ε, εντατικοποιηθούν και να μην σταματήσει η εφαρμογή τους. Και θα πρέπει να εξεταστεί και ο παράγων ε, ο διορθωτικός για τον άνθρακα. Δηλαδή σχέση που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών καυσίμων. Ας πούμε τα, το υγροποιημένο αέριο παράγει πολύ λιγότερα τέτοια καυσαέρια από ότι το, η κλασική βενζίνη και το πετρέλαιο. Και αυτός ο παράγοντας, ο διορθωτικός του άνθρακα θα πρέπει να εξεταστεί πιο προσεκτικά. Ε, πιστεύει ότι μπορούμε να βρούμε συμβιβασμό και όσον αφορά την αξιολόγηση για τον κύκλο ζωής που συζητούμε. Πολλές ομάδες υπέβαλαν τροπολογίες επ' αυτού και όπως προανέφερα Σήμερα δεν, δεν θέμα να φέρουμε σε δυσχερή θέση την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά θέλουμε να εξετάσουμε όλη την αλυσίδα ε, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην αξιολόγηση του κύκλου ζωής. Όσον αφορά τους τεθέντες στόχους, ο κύριος Σαλίνη είναι κάπως απογοητευμένος, διότι πολλές τροπολογίες και πολλά στοιχεία που συμπεριλαμβάνουν δεν έχουν συμπεριληφθεί στις συμβιβαστικές και περιμένει και ελπίζει ότι τα στοιχεία αυτά για το 2025 και για το 2030 θα τύχουν μεγαλύτερης προσοχής και συζητήσεως. Διότι είναι απαραίτητο να διεξαχθεί περαιτέρω συζήτηση από αυτόν. Ταυτόχρονα εκτιμά και το γεγονός ότι σε διάφορα, έχουν καθοριστεί διάφορα επίπεδα φιλόδοξων στόχων και γίνεται διάκριση μεταξύ των γιοταχή και των λεωφορείων και των μικρών φορτηγών και είναι καλό ότι αυτό ελήφθη υπόψη από την εισηγήτρια. Αυτά για την ώρα, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Βαντεκάπ. Κύριε Ζατόφσκι, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ο σκιώδης συγκητής, ο κ. Τσνόφσκι δεν είναι εδώ σήμερα και στη συγγνώμη γι' αυτό ε, διότι χθε το βράδυ βεβαίως ε, έλαβε χώρο ένας τρίλογος που κράτησε μέχρι πολύ αργά για την Ενεργειακή Ένωση. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρώτη σειρά τροπολογικών συμβιβασμών και θα ήθελα να αναφερθώ στα πιο σημαντικά ζητήματα για τους και εισηγητή το δικό μας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια διασύνδεση μεταξύ των στόχων που έχουν τεθεί για το 2025 και το 2030. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρώτο σημείο αναφοράς το 2025 πρέπει να είναι λιγότερο φιλόδοξο για να εξασφαλίσουμε ότι θα ακολουθήσουμε τον ορθό δρόμο για να πετύχουμε τους ρεαλιστικούς στόχους του 2030. Έτσι λοιπόν η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να είναι απαρέ... απαρέγκλητη για τους στόχους του 2025 και του 2030. Τελειώνοντας, να πω ότι και ο συγητής ε, θέλει να επιτευχθεί μια ισορροπημένη συμβαστική λύση με τον εισηγητή και τους λοιπούς συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ζατοφσκή. Ο κύριος ε, Ράντος έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε ε, και την Κομισιόν για την πρότασή τη που είναι αρκετά καλή, είναι ισορροπημένη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια θέση που είναι πολύ κοντά ε, στι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι αρχικέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά του στόχου του 2025 και του 2030, εμεί θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε και λίγο πιο φιλόδοξοι παραμένοντας βεβαίως ρεαλιστές μεταξύ των στόχων για το 2025 κατά τη γνώμη μας μπορούμε να συζητήσουμε ε, για το τι θα μπορούσε να γίνει το 2026 και το 2027 να τα πάμε λίγο πιο μετά ή να τους καταργήσουμε τους στόχους αυτούς στους ευρωπαϊκούς δρόμους υπάρχουν οχήματα τα οποία είναι παλαιότερα των 11 ετών προτείνουμε λοιπόν μια τροπολογία που να ενθαρρύνει την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα καύσιμα ε, με λιγότερη μόλυνση για να ενθαρρύνουμε αυτή τη χρήση και για οχήματα που δεν είναι καινούρια. Και προτείνουμε η παρακολούθηση ε, των καυσίμων και των εκπομπών να είναι διαθέσιμη ψηφιακά. Χαιρόμαστε που λήφθησαν υπόψη οι τροπολογίε μα από την εισηγητή και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή, Επιβάλλοντα βεβαίω και άλλε τροπολογίε. Ευχαριστώ τον κύριο Ράντο. Ο κύριο Μπασέτσκου έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ε, λέει ο κύριο Έκχαουτ, για την πρώτη σειρά συμβασμών. Τα είδαμε στην πρώτη συνεδρία των σκηνών εισηγητών, τα ξαναδούμε και στην επόμενη. Και εμείς ε, αναζητούμε συμβαστικές λύσεις και νομίζω ότι για μια σειρά ζητήματα σίγουρα μπορούμε να το πετύχουμε αυτό για τον κύκλο ανάλυση, τον κύκλο ζωή μάλλον και τη σχετική ανάλυση. Χαίρομαι που επιτέλου υπάρχει ευρεία υποστήριξη και να εξετάσουμε την ανάλυση του κύκλου ζωή ε, από όλου. Όταν συζητούσαμε τα βιοκάψιμα βέβαια, κανεί ε, δεν το ήθελε αυτό. Τώρα που συζητάμε ηλεκτρονικά οχήματα, ξαφνικά όλοι το θέλουν. Είναι συναρπαστικό. Ε, εν πάση περιπτώσει, εγώ το καλωσορίζω. Δεν θα κάνουμε βέβαια τον πλήρη κύκλο ζωή. Ε, εγώ αυτό θα ήθελα να, βάλουμε, να μιλήσουμε για πλήρη κύκλο ζωή. Ε, όχι μόνο όταν συζητούμε για τα οχήματα, αλλά και για τα βιοκαύσιμα και για όλε τι άλλε εναλλακτικέ. Τώρα για την τεχνολογική ουδετερότητα και εδώ ε, θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ε, πάλι όταν συζητούσαμε το βιοκαύσιμα πότε, ε, πότε μιλήσαμε για τεχνολογική ουδετερότητα. Μιλήσαμε για στόχους, υποστόχους, υποϊποστόχου και ξαφνικά τώρα θυμηθήκαμε την τεχνολογική ουδετερότητα. Δεν είμαστε και τόσο συνεπεί. δεν, είναι, δεν μας διακρίνει η συνέπεια, τουλάχιστον κάποιου από του συναδέλφου εδώ. Το πιο σημαντικό πάντως είναι το επίπεδο των στόχων. Ε, ε εκεί πρέπει να εργαστούμε ε, και βεβαίως εδώ δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχει και γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος πλέον που μιλάει για 50%. Γερμανικό Υπουργείο, έτσι. Ε, η Γερμανία δεν είναι τόσο φιλόδοξη ό,τι αφορά τους στόχους για τα αυτοκίνητα. Να λοιπόν όμω που ένα γερμανικό Υπουργείο στα 50%. όλο και περισσότερε χώρες λένε ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανεπαρκείς για να εφαρμοστούν οι συμφωνίε του Παρισίου και χθε όταν ο κ. Μακρόν και η κυρία Μέρκελ συναντήθηκαν είπαν πολλά για του πρόσφυγε, είπαν πολλά για το ευρώ, αλλά είπαν επίση ότι θεωρούν ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη ε, στην επόμενη COP24. Αυτό κάτι σημαίνει και για του διάφορου κλάδου. Όταν ο κ. Καμπ λέει ότι όλοι οι κλάδοι πρέπει να παίξουν τον ρόλο του και όχι μόνο αυτή η κοινοβιομηχανία η οποία τιμωρείται, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η μεταχείριση ε, έτσι, τιμωρητική για την αυτοκινητομηχανία στις προτάσει της Κομισιόν. Αντιθέτως, ε, ε, μάλλον να ανταμείβεται. Εάν δούμε όμως την εφαρμογή των Παρισίων και του στόχου που έχουμε θέσει, να έχετε κατά νου ότι το μέτρο το οποίο έχει μεγαλύτερη, την καλύτερη σχέση κόστου κόστος-οφέλους είναι να φτιάξουμε πιο αποτελεσματικά οχήματα στο να εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Έχουμε πολλά για το ETS, πολλά για, το, για, τη, γεωργία, για τη γεωργία, αλλά το λεξίδιο του άνθρακα και τα οχήματα είναι εκεί όπου η Ευρώπη μπορεί να πετύχει τα περισσότερα. Και είναι κρίσιμο αυτό για τις χώρες για να μπορέσουν να πετύχουν και τους εθνικούς τους στόχους ε, που προέρχονται από τον κανονισμό του διαμερισμού της προσπάθειας. Εάν λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό τώρα, οι χώρες, τα κράτη-μέλη δηλαδή, θα δυσκολευτούν να, πετύχουν τους εθνικούς στόχους ε, για το 2030. Διότι αν τα, ε, αυτή, η προσπάθεια δεν προκύψει από τι μεταφορέ, θα προκύψει από αλλού, από τη γεωργία παραδείγματο χάρη. Όσοι λοιπόν μιλάνε για το Παρίσι και για την εφαρμογή του και για την ε, ισόνομη, ισόνομη κατανομή, πρέπει να φτάσουν στο συμπέρασμα ότι οι προτάσει τη Κομισιόν για του στόχου είναι σαφώ ανεπαρκής, σαφώς ανεπαρκής. Ξέρω ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτό εδώ, διότι έχει, υπάρχει μια ιεραρχία. Καλό όμως είναι και η Κομισιόν να αλλάξει τη στάση της, διότι εάν αποτύχουμε εδώ, είναι βέβαιο ότι το κράτη-μέλη θα ακολουθήσουν ένα δρόμο εξαιρετικά, ένα αποτελεσματικό, εξαιρετικά κοστοβόρο. Ε, ακόμα και η Κομισιόν λέει ότι ο δικός χάτης ε, τον Νοέμβριο θα δείξει ότι οι στόχοι θα είναι υψηλότεροι. Σας παρακαλώ λοιπόν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργαστείτε ε, και ξαναδείτε το, ξέρω δεν, δεν μπορείτε να το κάνετε τώρα, πρέπει να περάσει, περάσετε από όλη τη συνηθισμένη διαδικασία, ελπίζουμε πάντως την επόμενη φορά να ακούσουμε κάτι άλλο από την Κομισιόν, είναι κάτι που το χρειαζόμαστε, πρέπει πραγματικά αυτός ο κλάδος να καθαρίσει πιο γρήγορα. Ευχαριστώ τον κύριο Έκχαουτ. Ε, θα περιορίσω, θα περιορίσω όμως το χρόνο, ιδάλλως ε, θα δυσκολευτούμε. Ο κύριος Ρικέ, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ναι, ναι, θα είμαι σύντομος. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα που θα, θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία, μια γενική συμφωνία. Οι δείκτες, ε, τους συστήματα μέτρηση και αξιολόγηση ε, για τον άνθρακα, για τι εκπομπέ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε από αυτόν. Είναι απαραίτητο να γίνουν διορθώσεις διότι υπήρξαν παραλήψεις. Ε, θέλω να πάω όμως στο εξή. Ο στόχος, δηλαδή η πρόταση της Κομισιόν το 15 και 30, κάποιοι λένε και 75, κάποιοι λένε και 100, αλλά αυτή η μείωση δεν θα γίνει ούτε μέσω της τεχνολογικής πρόοδου σε ό,τι αφορά τα θερμικά, ούτε μέσω των βιοκαυσίμων αλλά μέσω μιας, μετα... μιας αλλαγής, μετατροπής της αγοράς προς την κατασκευή οχημάτων με μηδενικές εκπομπές. Αυτό το πέρασμα όμως ε, στα αυτοκίνητα με μηδενική, ε, μηδενικές εκπομπές αφορά όλο τον κλάδο, τη βιομηχανία και όλες τις, και όλες τις σχετικές ε, ε, δραστηριότητες. Γιατί αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτές τις προτάσεις όπως αυτές που λένε οι πράσινοι, ουσιαστικά θα καταργήσουμε θα, θα διαρρέσουμε δια τριάμιση τις θέσεις εργασίας στην οικονομικανία. Δηλαδή μιλάμε για κάποια εκατομμύρια ανθρώπους. Και δεν θα υπάρξουν πωλήσει για αυτά τα οχήματα αν δεν λύσουμε τα προβλήματα με τι μπαταρίε, ε, τα προβλήματα τεχνολογικά, τα προβλήματα παραγωγή. Θα υπάρξουν και προβλήματα οικονομική υποστήριξη από τα κράτη-μέλη στην πώληση αυτών των οχημάτων. Ξέρουμε ότι όταν δεν τα υποστηρίζουμε δεν πολλούνται. Ε, και τέλο, θα, χα, θα χαθούν και κάποια ωφέλη σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν ότι εντάξει καλό είναι να έχουμε ένα στόχο, αλλά δεν πρέπει να φτάσουμε το στόχο αυτό όπω να είναι. Ε, ευχαριστώ κυρία Ντελμόντε. Η Ντελμόντε έχει το λόγο για 1,5 λεπτό και αυτή παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καταρχά, ευχαριστώ την συγγήτρια για την πρόταση. Ξέρουμε ότι ο τομέα των μεταφορών είναι ο κυριότερος υπεύθυνος σχετικά με τους δρύπους και τη μείωση, αλλά νομίζω θα πρέπει να διακρίνουμε τα γιοταχή από τα εμπορικά οχήματα. Και κάνω και μια έκκληση να μην σταματήσουμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί ο κόσμος των εμπορικών οχημάτων μας δείχνει ότι μπορεί να είμαστε πιο προχωρημένοι και να έχουμε εναλλακτικά καύσιμα, όπως το LNG. Βέβαια, αυτοί που Οφελούνται, πρέπει να κάνουν και κάποιες αξιολογήσεις για το κατά πόσο είναι σκόπιμο να εξοικονομούν χρήματα όσον αφορά τους εφοδιασμούς τους με καύσιμα. Η αυτονομία επίσης, η δυνατότητα φορτίου και βέβαια και το περιβάλλον όπου θα πρέπει να βάλουμε υπόψη μας το πλήρη κύκλο ζωής των οχημάτων. Να είμαστε λοιπόν φιλόδοξοι, αλλά να είμαστε ταυτόχρονα και συγκεκριμένοι ρεαλιστές και να μην χάνουμε την εστίασή μας. Δηλαδή θα πρέπει να ασχολούμαστε όχι μόνο με τα νέα οχήματα, αλλά, και με τα ήδη υπάρχοντα. Ωραία. Έχουμε τα νέα οχήματα που παράγονται, αλλά θα πρέπει να προσπαθούμε να μειώσουμε όλες τις εκπομπές. Αλλιώς θα έχουμε ένα αποτέλεσμα τελικό το οποίο δεν θα λύνει τα προβλήματα. Monsieur Ευχαριστώ κύριος Κράμερ, έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είπε ο κύριος Βαντενκάμπ ότι δεν πρέπει να τιμωρήσουμε την αυτοκρατομηχανία. Αυτοί μας τιμωρούν όμως, διότι είναι ο μόνος κλάδος όπου οι εκπομπές αυξάνονται. Εμείς έχουμε επενδύσει βεβαίως στους άλλους τομείς, αλλά Μα βυθίζει τελικά η μηχανία. Πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα. Στη Γερμανία προβλέπουν 5 δι για τα ηλεκτρονικά οχήματα, ε, τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Και θέλουμε να φτάσουμε σε αύξηση 50% ε, για τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Η κυρία Μέρκελ μας είπε χθε ότι αν δεν σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή θα, αυτό θα μας κοστίσει πολύ. Βέβαια, βεβαίω πάνε γρήγορα τα πράγματα στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ε, και τελικά τα φρενάραμε έτσι ώστε να υπάρχει μια ευκαιρία και για τον άνθρακα στο μέλλον. Ε, έτσι λοιπόν, ε, εμείς σκοτώνουμε εκατομμύρια, χιλιάδες ανθρώπους ε, με τις εκπομπές διοξείδου του άνθρακα, αλλά εξακολουθούμε να επιδοτούμε και τον δίζελ. έτσι. Ε, ξέρουμε από προέρχεται το ρεύμα, δεν προέρχεται από την πρίζα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το σύνολο του τη αλυσίδας παραγωγής. Ε, κύριε Ρικέ, η Ντέμλερ Benz πριν από 30 χρόνια γνώριζε ότι η αυτοκινητομηχανία θα είχε μέλλον μόνο αν υπάρχει κινητικότητα. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν φορτηγά, ε, τρένα που κουβαλούν φορτηγά και τώρα η Mercedes εξαρτάται μόνο από τα οχήματα, από τα ΙΟΤΑΧΗ. Ε, αν η Daimler είχε ακολουθήσει ε, την Ρόιτερ, τότε θα είχε μέλλον, θα είχε ένα μέλλον ρόδινο, ε, κατασκευάζοντας τρένα, αεροπλάνα κτλ. Αυτό πρέπει να κάνει η αυτοβιομηχανία, αλλιώς ε, θα αποτύχει και θα βαλτώσει, όπως οι ενεργειακές εταιρείες που τις ανανεώσιμες φυσικές ενέργεια τις αγνόησαν για χρόνια. Θα πρέπει να προσαρμοστεί. Ε, ευχαριστώ. Ναι, να απαντήσω λίγο εν συντομία στον συνάδελφο τον Μπάζ, ε, τον Μπάρτ μάλλον, ε, τον κύριο Έκχαουτ. Εμεί εμείς είμαστε υπέρ της βεβαίως, αλλά πρέπει να δούμε που προέρχεται η ενέργεια από μπαταρίες που παράγονται, ε, που έχουν ένα κόστος παραγωγής. Ε, πρέπει να υπάρχουν τα σημεία επίσης πρόσβασης. Ε, εμείς ζητήσαμε τεχνολογική ουδετερότητα και για τα βιοκαύσιμα. Θα πρέπει να δούμε επίσης και τις αναλλακτικές υποδομές. Είναι σημαντικό κατά τη φάση της εφαρμογής να μην σκεφτόμαστε μόνο την κινητικότητα, να σκεφτόμαστε το σύνολο των τρόπων με τους οποίους οι υποδομές θα βοηθήσουν και πρέπει να το κάνουμε αυτό από κοινού για να προχωρήσει η ατζέντα κατά της, της, Ε, λοιπόν, ο κύριος Άρθου Ράνκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στήσει το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Βεβαίω δεν μιλάω στο όνομά μου, μιλάω στο όνομα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Έκχαουτ ε, ε, ήδη αναφέρθηκε σε μένα, καλοσύνη του. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε υποβάλει μια ισορροπημένη πρόταση. Δεν εξετάζουμε μόνο το θέμα των εκπομπών ε, θερμοκηπίου και τη μείωσή τους, ε, αλλά και τι θα συμβεί στον καταναλωτή, στον πελάτη και πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε στις καινοτομίες. Σε γενικές γραμμές αυτή η πρόταση πιστεύω ότι θα πετύχει αποτελέσματα στη μελέτη αντικτύπου νομίζω ε, φαίνεται ότι θα πετύχουμε το 40% τον στόχο ε, τον οποίο θέσαμε στο Παρίσι, αυτό είναι σαφές και μπορούμε να το εξηγήσουμε ε, εκ νέου εφόσον χρειαστεί. Όταν μιλάμε όμως για το γενικότερο ερώτημα της φιλοδοξίας που πρέπει να έχουμε, βλέπουμε εμείς ότι χθε το βράδυ φτάσαμε σε μια συμφωνία από το 30% στο 32,5% ότι αφορά την ενεργειακή αποδοτική χρήση ενέργειας ε, και για τις ανανεώσιμες υπάρχει αύξηση 32 από το 27 υπάρχει λοιπόν ε, αυτή τη μια τάση που μας δείχνει ότι θα πάμε σίγουρα πάνω από το 40% αυτό που συμβαίνει με το, με τις είναι πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει ο κλάδος. Και αυτό έχει να κάνει και με την απασχόληση, διότι εάν κάνουμε αλλαγές πολύ γρήγορα και εξετάζουμε τους στόχους του 50 ε, και του 70% που δεν είχαμε κατά νου αρχικά στην αξιολόγηση που για να δούμε πόσο δραστικές θα είναι αυτές οι αλλαγές ε, τα πρώτα αποτελέσματα όμως μας λένε ότι μπορεί να είναι αρκετά δραστικές επιπτώσεις για τον κλάδο. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο ρυθμός των αλλαγών θα μπορέσει να είναι τέτοιος ε, που να μην έχει, υπάρξουν απώλειες. Από την άλλη τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική κινητικότητα, υπάρχουν πολλά κίνητρα στην πρόταση για το πέρασμα προς τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Αυτό σημαίνει ηλεκτρονική κινητικότητα. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα βεβαίως είναι το θέμα της παραγωγής ε, μπαταριών. Ε, πρέπει να έχουμε καταρχήν τέτοιου είδου παραγωγή στην Ευρώπη, διότι αυτό θα έχει και θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση. Από την άλλη, και βεβαίω και αυτό χρειάζεται επενδύσει και προγραμματισμό, και το 2030 είναι σε 12 χρόνια. Είναι ο ρυθμό λοιπόν τη αλλαγή που είναι σημαντικό. και υπάρχει συζήτηση για τις πρώτες ύλε. Βλέπουμε ήδη κάποιες από τις τιμές των πρώτων που αυξάνονται. Το κοβάλτιο είναι ένα παράδειγμα. Ε, εάν λοιπόν έχουμε υψηλότερους στόχους από την πρόταση της Κομισιόν, εμείς φοβούμεθα ότι αυτό θα οδηγήσει σε ε, προβλήματα ε, σε ό,τι αφορά την προσφορά και τη ζήτηση αυτών των πρώτων και αντί να μειωθούν οι, οι τιμές, κάτι που θα γινόταν με μια ομαλή μετάβαση, μπορεί να αυξηθούν και αυτό στη μεταβατική περίοδο ε, νομίζω ότι θα είναι εμπόδιο. Θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Εξετάζουμε κάποιες ποσοτικές πτυχές αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες ε, να έχουμε ακόμα κάποια αποτελέσματα ε, τα οποία θα μπορέσουμε να φέρουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο για να γίνει μια καλή συζήτηση τους επόμενους μήνες. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την εφαρμογή της είναι αρκετά απλή. Να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το γνωστό σύστημα με κάποιες βελτιώσεις βέβαια περνώντας ε, στην WLTP για να μην έχουμε τα μειονεκτήματα του παρελθόντος. Αυτό που μας ανησυχεί είναι εάν περιπλακούν πολύ τα πράγματα στην πρόταση δηλαδή ανάλυση κύκλου ζωής. Ε, Βέβαια σημαντικό στοιχείο, πρέπει να το δούμε. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει υποχρέωση για το κάθε όχημα. Να ξέρουμε δηλαδή ποιος είναι ο κύκλος ζωής του. Ο κύριος Εκχαουτ αναφέρθηκε προηγουμένως σε αυτό, ε, αναφέρθηκε στον συνολικό, στον πλήρη κύκλο ζωής του οχήματος. Αυτό όμως ε, σημαίνει πολλές απαιτήσει αναφοράς για τους ε, κατασκευαστές και δεν νομίζουμε ότι αυτό αιτιολογείται. Επίσης, ε, ακούμε ότι υπάρχει το θέμα της διόρθωσης ε, του άνθρακα και ότι αυτό θα δημιουργήσει μια περιπλοκή, θα δημιουργήσει ένα διπλό κανονισμό. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, είναι το τελευταίο που ήθελα να πω. Στις ανώσιμες πηγές συνέργειας έχουμε έναν στόχο για τα ε, καύσιμα ε, υπάρχει δηλαδή εκεί ένα κίνητρο. Γιατί λοιπόν να έχουμε μια διπλή επιδότηση και μια διπλή καταμέτρηση τελικά του τι πετυχαίνουμε. Ε, να το μετρήσουμε δηλαδή αυτό και ε, στο διοξείδιο του άνθρακα. Θα ήταν αντιπαραγωγικό. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν σε διοικητικό επίπεδο στην πρόταση, στην πρόταση αυτή. Και έτσι ολοκληρώνεται και η παρέμβασή μου. Θα συνεργαστούμε τι επόμενε εβδομάδε με τον εισηγητή και του κοιόδη εισηγητέ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση τη Κομισιόν. Δύο λεπτά, η κυρία Ρεονταλόν, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπω ότι μιλάμε εδώ για την αυτοκίνητο βιομηχανία, μιλάμε για τα καύσιμα, τα ηλεκτρικά οχήματα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε σφαιρικά. Γιατί είναι αλήθεια ότι για τους ρήπους πρέπει να μιλήσουμε σφαιρικά. Έχουμε τις συμφωνίες του Παρισιού που μας επιβάλλουν να μειώσουμε όλους τους δρύπους από όλες τις πηγές. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι όταν μιλάμε για τεχνολογική ουδετερότητα δεν μιλάμε μόνο για τα ηλεκτρικά γιατί μία από τις προτάσεις που έχουμε ώστε να πάμε σε μηδενικούς ρήπους, παρόλο που δεν είναι η μόνη πρόταση, γιατί έχουμε και το υδρογόνο, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί δεν βλέπω εδώ ή δεν πιστεύω εδώ ότι κάποιοι από εδώ εμάς στην Επιτροπή Μεταφορών είμαστε κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Όλοι προσπιζόμαστε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Δεν θέλουμε όμως η αυτοκίνητο βιομηχανία να υποχωρεί σε σχέση με ανταγωνισμό όπως ο κινητικός ανταγωνισμός που καλπάζει και κάνει τη μετάβασή της προς τρόπους που προτείνουμε με ναι, χαμηλότερο κόστος, λιγότερους ρήπου κτλ. Θέλουμε λοιπόν αυτή την βιομηχανική διάσταση να την ε, προασπίσουμε, όπως και την κοινωνική διάσταση με τις θέσει εργασία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είμαστε τελικά υπερβολικά φιλόδοξοι παρά τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την αυτοκίνητη βιομηχανία μα. αν την αφήσουμε σε ένα περιβάλλον όπου θα είναι λιγότερο ανταγωνιστική. Οπότε θεωρώ ότι οι ανάγκες και οι σκέψεις μας θα πρέπει να λαμβάνουν αυτά τα πράγματα πολύ σοβαρά. Για τα υπάρχοντα οχήματα που ανέφεραν διάφοροι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι θέλαμε αρχικά να απελάβουμε κάποιες προτάσεις στη γνωμοδότησή μας για το θέμα των υπαρχόντων οχημάτων αλλά μου εξηγήσαν ότι δεν ήταν αυτό το αντικείμενο της έκθεσης και κάθε φορά που εξετάζουμε τα θέματα ένα προς ένα και όχι σφαιρικά, τότε δεν καταλήγουμε σε καλά αποτελέσματα. Ενώ θα πρέπει πραγματικά σε σφαιρικό επίπεδο, γενικό επίπεδο να βρούμε, να πετύχουμε αποτελέσματα. Τώρα για τις φιλοδοξίες και τους στόχους, τι θέλουμε ακριβώς. Θέλουμε η αυτοκίνηση να είναι πιο ανταγωνιστική και λιγότερο ρηπαίνουσα με τεχνολογία εχμής ή αντίθετα θέλουμε επειδή ακριβώ ε, φοβόμαστε κάποιες φάσεις οι οποίες είναι βέβαια φιλόδοξες αλλά λιγότερο ε, δεσμευτικές θα οδηγήσουν σε υποχώρηση της ε, αυτοκινητομηχανίας μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά, γιατί θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας όταν τα ξανασυζητήσουμε στις 26 του Ιούνιου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος, κυρία Αργονταλόν. Υπενθυμίζω ότι στις 10 του Ιούλη θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα κατευθείαν στην ακροασή μας για την ψηφιοποίηση στον τομέα των μεταφορών. Je vais demander Θα ζητήσω από τους εμπειρογνώμονες να έρθουν εδώ να καθίσουν στο πάνελ. Mes chers collègues, je vais vous demander de prendre place. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Και οι νεόφυτοι, καλώς ορίσατε κι εσείς, καθίστε. Allez-y, n'ayez pas peur. Καθίστε, μη φοβάστε, καθίστε, καθίστε. Μην τρέπεστε. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη ακρόασή μας σε σχέση με την ψηφιοποίηση στον τομέα των μεταφορών. Η Επιτροπή λοιπόν των Μεταφορών αποφάσισε σήμερα να διοργανώσει αυτή την ακρόαση επειδή όπως ξέρετε η ψηφιοποίηση είναι όλο και πιο παρούσα στην καθημερινή μας ζωή και στις μεταφορές. Νομίζω ότι Όλοι έχουμε εμπειρία στις ψηφιοποίησεις σε αυτόν τον τομέα των μεταφορών, είτε όταν κοιτάμε τα ωράρια, είτε όταν με το GPS προσπαθούμε να εξυπηρετηθούμε. Μιλάμε για αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα, ψηφιοποίηση, μιλάμε για συνεπιβατισμό, μιλάμε για μεγάλες καινοτομίες που σε ένα άμεσο μέλλον θα φέρνουν μεγάλες ανατροπές στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τις μεταφορές και στον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε τις επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Με την ψηφιοποίηση λοιπόν όλων των υπηρεσιών των μεταφορών μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των μεταφορών, την εξυπηρέτηση των επιβατών και την ολοκλήρωση των μεταφορών. Στόχος εδώ της ακροασής μας ξεκάθαρα είναι να ακούσουμε τους εκπροσώπους ε, υψηλού επίπεδου από το τομέα των μεταφορών και τον τουρισμό σε σχέση με την ψηφιοποίηση για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σήμερα και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις που μας περιμένουν. Ιδιαίτερα όσον αφορά υπηρεσίες όπως οι κοινοφιλείς υπηρεσίες στις μεταφορές και πώς ακριβώς τις επηρεάζει η ψηφιοποίηση. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους στην Επιτροπή μας των Μεταφορών και σας καλώ βεβαίως να τηρήσετε τον χρόνο μιλία σας. Θα είμαι αμήλικτη, λέει η Πρόεδρος. Ο κάθε εισηγητής θα έχει στη διάθεσή του 5 λεπτά. Θα δώσω και στη συνέχεια το λόγο στους ε, βουλευτές για να θέσουν ερωτήσεις και παρατηρήσεις, αλλά καταρχάς, συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τους τους τέσσερις νικητές του βραβείου Startup ε, Prize, του βραβείου Startup για την κινητικότητα. Οι τέσσερις αυτές επιχειρήσεις που ανέφερε η Πρόεδρος οι οποίε εκπροσωπούν μια startup, μια νεόφυτη επιχείρηση και που θα μιλήσουν για τρία λεπτά ο καθένας από αυτούς τους νικητές. Και μετά ο κύριος ε, Πικέ ε, μπορεί να πει για τα δικά του και αυτός. Ευχαριστώ κύριε Πικέ. Και μετά θα ακούσουμε τους δύο τρεις διορθώνει πρόεδρος εμπειρογνώμονές μας και μετά θα επανέλθουμε σε εσά για την παρουσίαση των εργαλείων που προτείνεται. Εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν αμέσως με τον κύριο Κριστόφ Κλενέρ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Είστε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκής Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Ταξιδιωτικών. Πείτε μας λοιπόν πώς βλέπετε την ψηφιοποίηση στον τομέα σας. Έχετε πέντε λεπτά και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Έχετε το λόγο. Έχουμε και μετάδοση μέσω ίντερνετ. Σας ακούει λοιπόν και το διαδίκτυο και οι χρήστες του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν επιτρέπετε θα ήθελα να μιλήσω αγγλικά. Ευχαριστώ πάντως για την ε, πρόσκληση. Είμαι ο Κρίστοφ Κλένερ από την ΕΤΣΑ που λέγαμε προηγουμένως. Δύο λόγια σχέση με την ε, ομοσπονδία μας. Έχουμε επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, ανεξάρτητες δηλαδή από τις, από τις επιχειρήσεις μεταφορών ή από τις επιχειρήσεις καθαρά τις ε, τουριστικές. Εκπροσωπούμε διάφορα είδη ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ε, ταξιδιωτικά γραφεία, απλούς χρήστες, οι οποίοι κλείνουν τέλος πάντων ε, με ένα και μοναδικό ενίο τρόπο όλες αυτές τις υπηρεσίες με διαφάνεια και ταχύτητα. Η ψηφιοποίηση λοιπόν στον τομέα των μεταφορών είναι κάτι το οποίο ζήσαμε στο πετσί μας τα τελευταία 30-35 χρόνια και νομίζω ότι ήμασταν ένας από τους πρώτους τομείς οι οποίοι αγκαλιάσαμε την ε, ψηφιακή τεχνολογία πριν το ίντερνετ κιόλας το Computer Reservation System, το CRS, αν το θυμάστε, που ανάγεται στη δεκαετία του 70 και του 80, επέφερε μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αγοράζουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες οι χρήστες. Σήμερα θα επικεντρωθώ στον τομέα της αεροπλοείας, στις αεροπορικές, γιατί μετά από 30-35 χρόνια, όταν έχουμε μεσολαβήσει διάφορες τεχνολογικές επαναστάσεις, εμείς αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις, εμείς και οι χρήστες βέβαια, και θα ήθελα να κάνω κάνα δύο παρατηρήσεις σχετικά με αυτό, γιατί είναι κέρυες. Τι σημαίνει λοιπόν ανα, ανεξάρτητη κατανομή σε σχέση με τις αεροπορικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες και πώς αυτό ωφέλησε τους ε, χρήστες. Εμείς θέλαμε να υπάρχει μια διαφανής και ανοιχτή αγορά που ωφελήθηκε βέβαια από την ψηφιοποίηση και όπως ξέρετε όλοι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν το άνοιγμα της αγοράς των αερομεταφορών. Αλλά αυτό δεν θα είχε τα ωφέλη που έχει, αν δεν είχαμε μια ανοιχτή αγορά διανομής, το οποίο δίνει στις αεροπορικές εταιρείες δυνατότητα να ανταγωνιστούν με ίσους όρους και δίνει επίσης δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε σωστές πληροφορίες για να κάνουν τις σωστές επιλογές. Έχει θεσπίσει κάποιες δικλείδες η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει την διαφάνεια για τους χρήστες. Υπάρχει ο κώδικας διοντολογίας, υπάρχει 1008 και οι αεροπορικέ εταιρείε δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση, όπως και οι χρήστες δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη θέση για πρόσβαση σε υπηρεσίες αυτού του είδου. Είδους υπάρχουν όμως κάποια σύννεφα στον ορίζοντα. Οι μεγάλε αεροπορικέ όπως πολύ γνωρίζετε εδώ στην αίθουσα, παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες και συστηματικά κάνουν διακρίσεις καλά κατά α, πλατφορμών που δίνουν με διαφάνεια τη δυνατότητα επιλογής στους χρήστες. Εδώ έχουμε να κάνουμε τα εστία τα οποία δεν κλείνονται απευθεία από τους ταξιδιώτες και έχουμε επίσης και την επιβολή κάποιων εξόδων, επιπλέον εξόδων, τα οποία επιβάλλονται στους χρήστες που αγοράζουν ιστήρια εκτός ε, κυκλώματος ε, αεροπορικών εταιριών. Τι κάναμε λοιπόν, υποβάλαμε μια προσφυγή στην Κομισιόν. Η Κομισιόν τι κάνει, ε, κολλησιεργεί, εδώ και τρία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια ανασφάλεια δικαίου, ένα κενό νομοθετικό, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν διακρίσεις κατά των χρηστών που θέλουν να συγκρίνουν τιμές από τις αεροπορικές όσον αφορά αυτή την διανομή των υπηρεσιών. Οπότε η διαφάνεια εδώ απειλείται και τα επιτεύγματα της δεκαετίας του 90 που είχαμε το άνοιγμα αυτή τη αγορά έχουν τεθεί ένα αμφιβόλο. Εμείς λοιπόν καλούμε το Κοινοβούλιο ως συνομοθέτη να πιέσετε την Κομισιόν ώστε να εφαρμόσει σωστά τους κανόνες και να αξιολογήσει την συμπεριφορά συγκεκριμένων αεροπορικών για αυτά τα θέματα. Αυτό είναι ένα, ένα έδος ε, καθήκοντος πρέπει να θέσετε στην Κομισιόν και αυτή πρέπει να το λάβει υπόψη της σοβαρά. Η αναθεώρηση των κανόνων της ε, αεροπλοείας, των αερομεταφορών μάλλον, θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια και λαμβάνοντας πάτο υπόψη σοβαρά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των χρηστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με δεύτερο εμπειρογνώμα. Το κ. David Batchelor, υπεύθυνο διεθνή σχέσης εντός του ΣΕΖΑΡ, και υπεύθυνο για νέο χώρο ΕΦΗ e για τον καθαρό ατμοσφαιρικό ή καθαρή ατμοσφαιρικό αέρα και σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που δίνετε στη ΣΕΖΑΡ τη δυνατότητα να μιλήσει σήμερα στην κοινοπραξία. Θα πω μερικά λόγια για το θέμα γενικά και μετά θα μιλήσω για τα μη επανδρομένα επτάμενα οχήματα, τα drones και τον χώρο που ελέγχουμε. Να αναφερθώ στο ΣΕΖΑΡ. Είμαστε μια σύμπραξη ιδιωτικού τομέα, δημόσιου τομέα, δημιουργηθήκαμε το 2007. Ασχολούμεθα με το τεχνικό πυλώνα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και στόχος μας είναι να έχουμε συντονισμένη έρευνα και σχετικές δραστηριότητες, υποστήριξη της αγοράς ελέγχου ε, της κυκλοφορίας στην Ευρώπη και για τον εξυγχρονισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Eurocontrol μας δημιούργησαν για τον έλεγχο ενέργειας κυκλοφορίας και μαζί με 19 μέλη ε, έχουμε υπό την αιγίδα μας 100 εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συναθρίζουμε τους πόρους στην Ευρώπη για τον συγχρονισμό της διαχείρισης της ενέργειας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Γιατί μιλάμε για ψηφιοποίηση, βλέπουμε ότι το μέλλον των αεροπορικών μεταφορών θα είναι δραματικά διαφορετικό από το παρελθόν. Πέρα από τη μεγάλη ανάπτυξη στις παραδοσιακές, παραδοσιακές αερομεταφορές που βλέπονται και νέους χρήστες θα έχουμε όσον αφορά τους εθέρες και μεγάλη εκεί, ε, μεγάλοι λόγοι γι' αυτό. Έχουμε περισσότερο πληθυσμό θα ζει σε πόλεις, αύξηση του πληθυσμού, άρα θα έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες κινητικότητας στον αστικό τομέα θα έχουμε ταχεία εξέλιξη τεχνολογία, κυρίως όσον αφορά το αυτοματισμό, τεχνητή νοημοσύνη, εκμάθηση ε, των μηχανών σε γνώσεις και θα είναι η εθέρες στο μέλλον. Αντί να έχουμε χιλιάδε αεροσκάφη θα πετούν ταυτόχρονα όπω σήμερα, μπορεί να έχουμε εκατοντάδε χιλιάδε υπτάμενα οχήματα που θα είναι διασυνδεμένα και θα ύπτανται. Μέσω του ΣΕΖΑΡ εστιαζόμεθα επί των τεχνολογικών δομικών υλικών για την κατασκευή του συστήματος Σεζαρένα. Είχαμε 63 λύσεις που βρήκαμε, που συνοψίζονται στις, στον κατάλογο με λύσεις Σεζάρ και με το πρόγραμμα Σεζάρ 2020 έχουν πάνω 60 προγράμματα που έχουν δρομολογηθεί διερευνητική έρευνα, βιομηχανική έρευνα και επιδείξεις μεγάλης κλίμακας και πολλά από αυτά τα προγράμματα αφορούν την ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση είναι ένα ευρύ όρο, καλύπτει πολυσχηδεί δραστηριότητε, δεν θα σε λεπτομέρειε. Ουσιαστικά Έχουμε αυτόνομα οχήματα, μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, ε, εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, οι υπηρεσίε δεν χρειάζεται να. Ε, οι παρέχονται κοντά στον ενέργειο χώρο που εξυπηρετούν. Τα big data, ανάλυση των big data, κυβερνοασφάλεια. Όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία της ψηφιοποίησης των αεροπορικών μεταφορών. Στρεφόμενος προς τα drones, είναι σαφές ότι η αγορά των μη παντρωμένων υπταμένων οχημάτων αναπτύσσεται τάχιστα, προσφέρει νέα ωφέλη οικονομικά και κοινωνικά και γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός για τι μεταφορές έχει σαν στόχο τα drones να ενταχθούν στον ευρωπαϊκό ενέργειο χώρο σε φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα να ενταχθούν αρχές ε, του 2019. Πέρσι η κοινοπραξία Σεζάρ έδωσε, ετοίμασε χώρο για ένα νέο πρόγραμμα για διαχείριση του εναρίου χώρου για τα drones. Εκεί έχουμε μεγάλο ποσοστό ψηφιοποίησης και αυτόματες λειτουργίες και με την πάρα του χρόνου όλα αυτά θα στηρίξουν αποτελεσματική και ασφαλή πρόσβαση στον ενέργειο χώρο μας για μεγάλο αριθμό μη επανδρομένων διδαμένων οχημάτων διαφόρων ειδών. Οπότε το U-Space παρέχει ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει στο μέλλον οι εσδήποτε απλές αποστολές συμπεραβαμένων και πτυχών που θα αφορούν την αστική κινητικότητα, όπως ελπίζουμε. Λοιπόν, τιμάσαμε αυτό το σχέδιο, το αρχικό. Εκεί εντοπίσαμε σταδιακή ε, εισαγωγή των νέων υπηρεσιών με μεγαλύτερο αυτοματισμό και διασυνδεσιμότητα από U1 μέχρι U4 είναι οι κατηγορίες που δημιουργήσαμε. Το U1 είναι βασικές ε, υπηρεσίες που ελπίζουμε να λειτουργούν μέχρι του χρόνου. Και μετά ξεκινάμε με διάφορα διερευνητικά επιστημονικά προγράμματα μαζί με την ΕΑΣΑ ε, και αργότερα στο έτος ξεκινάμε διάφορες επιδειξεις για να στηρίξουμε τις υπηρεσίες EU2 που θα ε, εφαρμοστούν στο μέλλον. Περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν συνολικά για την υποστήριξη αυτών των ερευνητικών ε, δραστηριοτήτων και των επιδείξεων ρυθμό καινοτομία επιταχύνεται. Είναι σαφέ. Αυτό είναι πρόβλημα βέβαια για το μέτρο μεταφορών, διότι ε, η νέα τεχνολογία χρησιμοποιείται με αργού ρυθμού όσον την ασφάλεια. Εμεί έχουμε επιταχύνει σαν Caesar την καινοτομία. Ε, λοιπόν, η ψηφιοποίηση προχωρά, η ασφάλεια είναι πολύ βασικό παράγον όσον αφορά τα συστήματα αεροπλοεία στο μέλλον και η κοινοπραξία του Σέζαρ είναι το όχημα για την ψηφιοποίηση των αερομεταφορών στο μέλλον. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για αυτή την παρουσίαση, κυρίως για τους στόχους και που εστιάζει το πρόγραμμα Σέζαρ. Και τώρα στρέφομαι προς τον κύριο Γκαέλ Μουσκέ. Ένας από τους εμπειρογνώμονες είναι των διασυνδεδεμένων οχημάτων και των open source του ανοιχτού λογισμικού. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Οπότε καταπολεμείτε, είσαστε, διδίσατε αυτό το φορέα που καταπολεμά, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των φυσικών καταστροφών. θα σας ακούσουμε μεγάλη προσοχή, διότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Ευπρόσδεκτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας. Πρόεδρος μιας ένωσης που έχει σαν στόχο για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση με ευχαρίστηση, διότι καλύτερο τρόπο για να δοκιμάσουμε το μέλλον και το πώ θα εξελιχθούν οι μεταφορέ είναι να, το πώ θα αντιμετωπίζονται φυσικέ καταστροφέ οι μεγάλε. Αυτό κάνουμε σε απομακρυσμένε περιοχέ. Εγώ γεννήθηκα στη Γουαδελούπη και τακτικά κάνουμε ασκήσει για το τσουνάμι ε, δοκιμάζουμε κάποιους μηχανισμούς ραδιοφωνικούς, ε, ερασιτέχνες ε, που θέλουν όλοι αυτοί που έχουν τεχνικά μέσα για κοινοφελείς σκοπούς να διαθέσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους. Θέλουμε να έχουμε τέσσερις πυλώνες καινοτομία ψηφιακής. Το open source καταρχάς, τα open data είναι το δεύτερο, open standards και open hardware είναι τέσσερις πυλώνες. Open data λοιπόν είναι υποχρέωση σε πολλές χώρες και σε περιφερειές να διατίθενται τα στοιχεία που παράγονται δημοσίως και πολίτες που παράγουν τα στοιχεία να τα παρέχουν. Έχουμε το Open Street Map. Ξέρετε τι είναι το Open Street Map. Καταλαβαίνετε τι είναι. Ωραία. Για εκείνους που δεν το καταλαβαίνουν, είναι ένα πρόγραμμα που γεννήθηκε στην Ευρώπη, στην Αγγλία, Wikipedia χαρτογραφική είναι ουσιαστικά. Έχει πολλούς χρήστες. Χαρτογραφούν τις πόλεις τους, τις πρωτεύουσές τους, τη χώρα τους, ε, ε, τα δίκτυα των μεταφορών και ε, τουριστικούς τόπους και έχει παράξει αυτό το πρόγραμμα πάρα πολλά στοιχεία, τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και είναι ένα από τους καλύτερους φορείς σήμερα καινοτομία στις μεταφορές. Δεν θα υπάρξει καινοτομία κυριαρχία, αν θέλετε, ανεξαρτησία και θετική εξέλιξη, αν αυτά τα στοιχεία παραμείνουν ε, ιδιοκτησία των επιχειρήσεων που έχουν το μονοπόλιο και που ε, τιμολογούν την πρόσβαση σε αυτά τα ψηφιακά στοιχεία χαρτογράφησης. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις μας, οι χώρες μας να παράξουν στοιχεία για ελεύθερη χαρτογράφηση όπως το OpenStreetMap που δίνει ελεύθερα τα στοιχεία, ανοιχτά, δωρεάν, τυποποιημένα χαρτογραφικά στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν χρειάζεται να επανακαθορίσουμε τα πρότυπα, τα χαρτογραφικά SAE. Το open source, δεύτερο πυλώνα, ελεύθερο, το ανοιχτό λογισμικό, ένα φορέα καινοτομία. Έχουμε πολλέ εταιρείε που έχουν δεσμευθεί και πολίτε να παράξουν αυτά τα στοιχεία και αυτά τα ελεύθερα, τα ανοιχτά λογισμικά. Η SNCF στην ε, Γαλλία χρησιμοποιεί το OpenStreetMap μέσω διαφόρων ειδών λογισμικού για να δίνει σε πραγματικό χρόνο που βρίσκονται τα τρένα ή να δίνει πληροφορίε στου ταξιδιώτε. Πάρα πολλά προγράμματα υπάρχουν ανοιχτή πηγή, open source, όπω Automotive Linux για τους ε, πολίτες που θέλουν να δίνουν στοιχεία και λογισμικό που επιτρέπει στους οδηγούς στους οδηγούς να έχουν ψηφιακές ε, υπηρεσίες που βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους. Το open standard, τα ελεύθερα πρότυπα, υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα. Μιλήσαμε για αυτά της αεροπλοείας, το IS. Οι αναμεταδότες των σκαφών που σε πραγματικό χρόνο δίνουν στοιχεία συνεχώς, τα ωράρια, των δρομολογίων, των τρένων, των τραμ, των λεωφορείων, όλα αυτά τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται είναι πολύ σημαντικά διότι ο καθένας μπορεί να αποφεληθεί, να έχει την ίδια δυνατότητα να έχει πρόσβαση στα μεταφορικά αυτά τα στοιχεία και να μπορεί έτσι να παράγει καινοτομία. Open hardware. Να παράγεται υλικό, είναι να παράγεται προϊόν, συσκευή που επιτρέπει ε, να έχεις διαδραστική επαφή, να, αυξάς, να αυξήσεις τα συστήματα ασφαλείας, ε, την ασφάλεια των συστήματων πληροφοριών. Είναι μια δίωδος αυτή, ε, μάλλον είναι μια βαλβίδα εδώ αυτοκινήτου. Από το 2012 υπάρχει αυτός ο μηχανισμός για να βλέπει κανείς την πίεση στα ελαστικά και τη θερμοκρασία των ελαστικών. Είναι υποχρέωση, αλλά δυστυχώ τα στοιχεία δεν είναι ψηφιακά. Ε, τότε, όταν θεσπίστηκε ο νόμος, δεν είχαμε φανταστεί πόσο ευάλωτο θα ήταν το αποτέλεσμα αυτού του εργαλείου που χρησιμοποιείται. Εμεί θα, θα πρέπει να το αποδείξουμε σαν πολίτε ότι μπορεί να έχει κάποια αποτελέσματα ένα ε, νόμο και να υπονομεύει την ιδιωτικότητα τη ζωή κάποιου, αν χρησιμοποιείται κακώ ε, μια συσκευή. Σαν πολίτε ε, έχουμε το δικαίωμα του πειραματισμού, όπω οι ραδιορεσιτέχνε. Έφερα μαζί μου αυτό το ραδιόφωνο, αν θέλετε, αυτό το μπομπό, διότι έχουμε και εμεί κάτι να πούμε στην καινοτομία σαν πολίτε. Δεν είμαστε απλοί πολίτε, είμαστε τεχνικοί, μηχανικοί, hackers. Η καινοτομία δεν είναι μονοπόλιο των εταιριών ή των μεγάλων ε, κρατικών εταιριών. Εμείς σαν πολίτες έχουμε λόγο όσον αφορά ε, διάφορα, διάφορες εταιρείες και ενώσεις ερασιτεχνών, ε, ράδιο ερασιτεχνών που εργάζονται στα πλαίσια της καινοτομία και προσπαθούν να συνεργαστούν με το τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Μισκέ, κύριε Μισκέ. Αυτοί ήταν οι τρεις ομιλητές που μας έδωσαν κάποιες ιδέες. Να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Θα ακούσετε δηλαδή τα ερωτήματα των μελών μας. Κύριε Βάντενκαμ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Κύριε Κλένερ, το ΕΛΚ στο παρελθόν είχε θέσει κάποια ερωτήματα για το θέμα αυτό, προφορικά ερωτήματα, η κυρία Μοντέρο πιο συγκεκριμένα, και είδαμε και η κυρία Μπούλ στην Επίτροπο, και το ερώτημα είναι το εξής Γνωρίζω βέβαια την απάντηση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τελικά κάτι γι' αυτό ή συνεχίζετε να λέτε ότι όλα είναι μια χαρά. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο, η διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως είμαστε πολύ αργοί. Οι Κινέζοι, παραδείγματο χάρη, είναι πολύ πιο γρήγοροι. Στι ΗΠΑ είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα αυτή τη στιγμή, βέβαια, ε, με τον κύριο Τραμπ, αλλά και εκεί παίρνουν τι αποφάσει πιο γρήγορα. Και εμεί έχουμε τι 28 χώρε με 28 κοινοβούλια ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βέβαια. και δυσκολευόμαστε να προχωρήσουμε. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το ρυθμό και τι θα κάνουμε γι' αυτό. Και ένα ερώτημα, ένα σχόλιο προς τον κύριο Μισκέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Διότι κάποιοι που κάποτε θεωρούσαν εγκληματίε, τώρα αποτελούν μέρο ε, του, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην πραγματικότητα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι παρκώ εμπειρογνώμονο για να μιλήσω για το hacking, αλλά χαίρομαι που είστε εδώ μαζί μα και ε, συμμετέχετε κι εσείς. Ε, ναι, όπως και να το κάνουμε, έχει ένα νέο καθεστώς. Ο κύρι, η κυρία Φώστερ έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που έχασα την πρώτη ομιλία. Είχα μια δουλειά. Δεν μπορώ να ρωτήσω και ερωτήματα. Ο τρίτος ομιλητής πραγματικά ήταν συναρπαστικά αυτό που ακούσαμε. Ε, βλέπουμε ταινίε με, τα, με τους hacker οι οποίοι χακάρουν τα μεγάλα συστήματα, τους κυνηγάει το FBI και τους πιάνει. Ε, αλλά γιατί δεν τους ε, προσλαμβάνει, διότι ε, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα έτσι. Είναι πραγματικά συναρπαστική αυτή η παρουσίαση. Τώρα για τον David Batchelor, χαίρομαι που τον βλέπω και βεβαίως ε, ήμουν εισηγήτρια ε, σε ό,τι αφορά την Σέζαρ. Είχαμε μια πολύ καλή επίσκεψη στην Ιάσο. Είχαμε μια συζήτηση με τον Πάτρικ Χίλ και, τους, ε, και το επιτελείο του. Ξέρω ότι η Ιάσο έχει το, το έγγραφο, το πρωτότυπο. Ξέρω ότι ε, πήρε χρόνο για να φτάσουμε στα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του βασικού κανονισμού. Δεν θα μιλήσω λοιπόν γι' αυτό, αλλά ω εισηγήτρια για την έκθεση για τα drones, για τα μη επανδρομένα, θα ήθελα να ξέρω τελικά πώ θα αποκινούμαστε. Δεν είμαι και τόσο ικανοποιημένη με την καθυστέρηση, ε, με το χρόνο που έχει χαθεί για να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Αυτό που γνωρίζω όμω είναι ότι υπάρχει κάτι σχετικά με το ελεγχόμενο ε, αέριο χώρο ε, σε ό,τι αφορά τα drones. Δηλαδή πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Το αφήνουμε δηλαδή στα κράτη-μέλη ε, να καθορίσουν τους κανόνες για τα drones. Το οποίο δεν είναι πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να δοθεί μια όθηση, διότι εσείς συνεργάζεστε μόνο με το ΣΕΖΑΡ οι Υπηρεσίε με τη διαχείριση σενάριου χώρου κάνουν τη δουλειά του. ε, ο καθένας προχωράει όσο πιο γρήγορα μπορεί, αλλά έως τώρα είχαν τα χέρια του δεμένα στο ΣΥΖΑΡ. Δεν ξέρω αν έχετε εσεί κάποια λύση να προτείνετε για να προχωρήσουμε, διότι είναι κρίσιμο το θέμα και είναι πολλά ε, τα πλεονεκτήματα για την Ευρώπη στην προκειμένη περίπτωση. Η κυρία Μάισνερ έχει τώρα το λόγο. Ναι, ευχαριστώ να ευχαριστήσω και τους ομιλητές. Δεν έχω ερώτημα για τον κύριο Κλάινερ. Χάρηκα που άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Μπάτσελορ, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Φώστερ, ε, εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα του ευρωπαϊκού ουρανού Εφόσον έχετε ήδη κάποια σχέδια σε επίπεδο ψηφιοποίηση ε, του ETM και θέλετε να, επι, να, να, εφαρμόσετε, να μάλλον να συμμετάσχουν, να εμπλακούν εδώ και τα drones, ίσως να είναι κάπως πρόημο αυτό, αλλά πιστεύετε ότι μπορείτε να βελτιώσετε την κατάσταση ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό ουρανό, διότι εάν η, η πλήρη ψηφιοποίηση ε, επέλθει, δεν ξέρω αν θα υπάρξει απαραίτητα και καλύτερη λειτουργία και πόσοι από εμά θα χρειαστεί να κάνουν παρακάμψεις στις πτήσεις τους λόγω των περιορισμών. Λοιπόν, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και τρίτη ομιλία. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που είπατε. Ήταν πολύ καλό το Open Suite Map στο οποίο αναφερθήκατε και μιλάτε για την προστασία των δεδομένων. Αυτός ο χάτης θα είναι δωρεάν. Έτσι, πληρώνει κανείς με τα δεδομένα του δηλαδή. Μπορείτε να μας εξασφαλίσετε όμως ότι εσείς είστε καλοί και άλλοι είναι κακοί. Διότι φοβάμαι ότι τελικά θα εξαρτώμεθα από τις επιχειρήσεις. Εμένα με ενδιαφέρει πρόοδο στο διαδίκτυο, αλλά πρέπει να υπάρχει επαστασία των δεδομένων. Πώς μπορείτε δηλαδή να επιλύσετε το θέμα αυτό, πώς μπορείτε να μας εξασφαλίσετε ότι σε εσά ε, τα δεδομένα αυτά θα είναι ασφαλή και όχι αλλού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόρ έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Κλέινερ. Αναφερθήκατε στο, στις υπηρεσίες της εναέριες. Εγώ είμαι υπέρ της ε, διαδικής μεταφοράς. Έχω κάνει και μια σχετική έκθεση. Λέω ότι πρέπει να μπορεί κάποιος με ένα μόνο εισιτήριο να μπορεί να πάρει το τρένο και το αεροπλάνο και το ταξί. Ε, πιστεύετε ότι η αγορά θα προσαρμοστεί στη ζήτηση ή πρέπει να υπάρξει ρύθμιση. Έχουμε αφήσει τα χέρια ελεύθερα στην αγορά και είπαμε ότι αν δεν γίνει τίποτα στο 2020 θα υπάρξει κανονισμό. Εσεί πιστεύετε ότι θα χρειαστεί κανονισμό. Η κυρία Μπίρκενεν έχει το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Όπως γνωρίζετε, το θέμα αυτό είναι σημαντικό για μας, ειδικά τα τελευταία έτη. Η ψηφιοποίηση στον τομέα των μεταφορών ε, είναι μια τάση έντονη. Όπως είπε ο κ. Βαντερκάμπ όμως, ε, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια μεταξύ κρατών μελών και θέλει χρόνο όσο το φτάσουμε σε μια νέα ψηφιακή αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από όλους τους εμπειρογνώμονες εδώ πώς το βλέπετε εσείς. Ε, ποια είναι τα πιο σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν ε, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ε, ε, και τις καινοτομίες στον δικό σας τομέα για την ψηφιοποίηση. Κανονισμός, ρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις ή τροποποιήσεις κάποιων κανονισμών που είναι επαπαλαιωμένοι ή κάτι άλλο. Να επενδύσουμε στην έρευνα, σε κάποιες δεξιότητες. Πώς το βλέπετε εσείς. Ποια είναι τα πιο σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δώσουμε μια όθηση στις, ε, στην καινοτομία και στις επενδύσεις στον τομέα της ψηφιοποίησης. Μάλιστα. Ευχαριστώ την κυρία Μπυρκέιν. να δώσω τώρα ξανά το λόγο στους ομιλητές μας μετά τις ερωτήσεις. Έχω και εγώ ένα ερώτημα για το πρόγραμμα U-Space. Θα ήθελα να ξέρω εάν οι ψηφιακές υποδομές ε, υπάρχουσες για τα πειράματα ε, εφόσον αυτές ε, ε, αναπτυχθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, ποιε θα είναι οι ανάγκε, ποιε θα είναι οι ανάγκε σε επίπεδο υποδομών, ψηφιακών υποδομών και ποιο ρόλο θα πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση αυτή, διότι όπω ξέρετε αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαπραγμάτευση για τα ζητήματα τα δημοσιονομικά. Και με τον κύριο Μισκέ το ερώτημά μου τι αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα ζητήματα των ε, δεδομένων που είναι στην καρδιά ε, της πρόκλησης για τον 21ο αιώνα. Λοιπόν, ο κύριος Μισκέ πρώτος, ή να πάμε ανάποδα, ή ο κ. μισκε πρωτος Κλέναρ πρώτα. Ο κ. κλεναρ Μισκέ, ο κ. μισκε ο κ. μισκε Ναι, ακούστε, ε, είναι ενδιαφέρον ε, να δει κανείς πώς καταλαβαίνει κανείς τον λέξη hacker. Μιλάμε συχνά για τους κακούς hacker. Οι περισσότεροι hacker όμως είναι καλοί. Είναι πλευρά των καλών για να το πω έτσι. Είναι άντρες, γυναίκες οι οποίοι αμφιβάλλουν, αμφισβητούν τα συστήματα όποια αν είναι αυτά. Ο στόχος μας είναι μελετώντας τα συστήματα αυτά να καταλάβουμε πώς λειτουργούν πρώτον, να τα καταστήσουμε πιο ασφαλή και ενδεχομένως για να τα ε, αλλάξουμε τη χρήση τους. Αυτή είναι η βάση της δουλειάς του hacker. Και να, να απαντήσω στα ερωτήματά σας για την ασφάλεια. Εδώ έχω ένα παράσημο από τις αερομετά, τις, ε, ε, την, αεροπορία στρατιωτική. Γνωρίζουν οι ενόπλες δυνάμεις ότι μπορεί να είναι χρήσιμα αυτά που κάνουμε για την υπεράσπιση, την άμυνα της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης εκεί σε αυτήν την αεροπορική βάση είμαι υπεύθυνο για ένα σχέδιο καινοτομία που εποπτεύει την ενέργεια κυκλοφορία. Θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες, ε, κάποια κλειδιά TNT από αυτά που μας επιτρέπουν να έχουμε ψηφιακή τηλεόραση δηλαδή ε, για να μπορούμε να παρακολουθούμε τα, όχι, τα αεροπλάνα, τα πλοία και τις πληροφορίες που εκπέμπουν. Αύριο θα είναι και τα drones και γίνεται και μια συζήτηση και για τους δορυφόρους, διότι και εκεί πρέπει να υποπτεύουμε τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με αυτούς τους στρατιώτες, τους στρατιωτικούς ως πολίτης για να δείξουμε πώς εμείς οι πολίτες, εμείς οι hacker ε, μπορούμε να βοηθήσουμε για μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη καινοτομία. Κλείνω την παρένθεση αυτή σε ό,τι αφορά τον ορισμό του hacker. Θα σα δείχνω απλώ ότι μπορεί να είμαστε από τη σωστή πλευρά εμεί οι hacker την πλευρά των καλών και να δώσουμε στοιχεία για την επικοινωνία, την καινοτομία, για αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερα. Τι μας περιμένει αυτό το καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη. Πυρκαγιές στο νότο της Γαλλίας, στο νότο της Ευρώπης γενικότερα. Θα πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθούμε, να εποπτεύουμε την αέρια κυκλοφορία για τα Καναντέρ. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή επαρκείς πόρους ε, ανθρώπινους ε, αλλά και οικονομικούς για να γίνει αυτή η δουλειά. Με διάφορες λοιπόν υπηρεσίες πυροσβεστικής, με τις, ένοπλε δυνάμεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε πληροφορίες όσο γίνεται περισσότερες αυτές τις ε, ε, δυνάμεις. Θα είμαι στην Μασαλία και μετά στην Κορσική την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε από κοινού να βρούμε ε, λύσεις, λύσεις για τις μεταφορές, ε, τις αέριες μεταφορές, αλλά και θαλάσσιες. Και τώρα για το OpenStreetMap, η καλύτερη εγγύηση ε, είναι ότι αυτές, αυτά τα δεδομένα πρέπει να είναι βεβαίως ποιοτικά, να σέβονται την ιδιωτική ζωή του καθένα ε, και να είναι ανοιχτέ σε όλους. Είμαστε διαφανείς. Ε, συμμετέχουμε σε πολλές ομάδες σκέψης, συνεργαζόμαστε και με την SNCF, από τους μεγαλύτερους μεταφορείς σιδηροδρόμων και η ποιότητα αυτών των δεδομένων, η ποιότητα και των εταιριών που δουλεύουν περί των δεδομένων αυτών μας επέτρεψαν στην SNCF να μας, να μας εμπιστευτεί και να χρησιμοποιούν δεδομένα αυτά ε, τώρα για τα γρήγορα τρένα. Ε, για τα open data γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που ήθελα, θα ήθελα, ε, πέρυσι σε μια διάσκεψη το είχα πει, αυτό που θα ήθελα και θα θέλαμε και άλλοι, είναι να είστε όσο γίνεται πιο κοντά στο τι συμβαίνει επί τόπου. Κοντά στους ανθρώπους αυτούς, άντρες, γυναίκες, ε, τους στρατιώτες, αυτοί που ε, προσπαθούν να σταματήσουν πυρκαγιές. Θα γίνει και μια ε, τέτοια άσκηση στις 5 Σεπτεμβρίου στη Ρεωνιόν ε, με μια προσωμείωση τσουνάμι που θα φορά το σύνολο του ωκεανού είναι μια ευκαιρία να έρθετε εκεί να δείτε επιτόπου πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα πώς εμείς ως πολίτες μπορούμε να αναβλώσουμε αεροπλάνα, να βλώσουμε μη επανδρομένα, drones, ε, κάνουμε βαθιμετρικές μελέτες. Ε, αυτά τα δεδομένα συνέχεια είναι στη διάθεση όλων. Θέλουμε λοιπόν να είστε εκεί επί τόπου για να δείτε πώς αυτοί οι κανονισμοί μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα και έτσι ώστε στην εφαρμογή τους ε, να είναι όσο γίνεται λιγότερο πεπαλαιωμένοι και να είναι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένοι και σε σχέση με την πραγματικότητα. Ευχαριστώ τον Γκάιλ Μισκέ. Δεν ξέρω εάν θα είμαστε ελεύθεροι 5 Σεπτεμβρίου, θα το ψάξουμε πάντως, θα δούμε αν μπορούμε να έρθουμε στη Ριουνιόν. Έχετε το λόγο κύριε Μπάτσελορ. Um, so Ευχαριστώ. Κάποια ερωτήματα υπήρξαν για το κατά πόσο καθυστερούμε στην Ευρώπη. Τα drones και η ολοκλήρωσή του, η ένταξή του είναι μια μεγάλη πρόκληση. Παγκοσμίω, πολλέ χώρε αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση για το θέμα αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά. Έρευνα και ανάπτυξη πρώτα, γιατί δεν ξέρουμε τι τεχνολογία χρειαζόμαστε και πώς θα πάνε τα πράγματα. Οπότε έρευνα και ανάπτυξη πρώτα και αφού έχουμε εκεί αποτελέσματα, μετά μπορούμε να θέσουμε τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς και όλα αυτά που θα επιτρέψουν να εφαρμοστούν αυτές οι προσπάθειες. Αναβήμα λοιπόν θα προχωρήσουμε, βήμα προς μήμα μάλλον, και βέβαια ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη πίεση από τη βιομηχανία, γιατί υπάρχουν μεγάλο ωφέλη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου θέλουν ήδη να προχωρήσουν γρήγορα οι βιομηχανίες. Και μάλιστα, μια και αναφέρατε και την Κίνα, είχα πάει εκεί πριν δύο εβδομάδε σε ένα εργαστήριο για τα drones. Και εκεί πραγματικά προχωράνε μπροστά. Ακόμα όμως δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο Αντιμετωπίζουν λοιπόν διαφορετική πρόκληση εκεί. Δηλαδή ακόμα θα πρέπει να αναπτύξουν το κανονιστικό πλαίσιο. Ακόμα δεν ξέρουν πώς θα είναι αυτό. Στη ΣΥΠΑ ήμουν εκεί τέσσερα χρόνια εκπροσωπώντας το ΣΕΖΑΡ ε, δουλεύοντα πάνω στην διαλειτουργικότητα τη επόμενη γενιά. Έχουν, τις επόμενες έχουν προχωρήσει και είπα έχουν συστήματα προχωρημένα, ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση που έχουμε κι εμείς. Και θα ήταν σωστό να πούμε ότι μάλλον δεν είναι και τόσο περισσότερο προχωρημένοι από εμάς. Ταυτόχρονα μαθαίνει ο ένας ε, από τον άλλον, γιατί έχουμε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας. Και μέσω και της ΙΚΑΟ ε, συνεργαζόμαστε, γιατί πρέπει να έχουμε συμβατά συστήματα. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν χρόνο και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε τη δουλειά μας στο ΣΕΖΑΡ. Ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη του πλαισίου του νομοθετικού και αυτά από μένα ενημερωτικά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος στόχος του ΣΕΖΑΡ αφορά τεχνολογίες και τα παραδοτέα Τώρα, η χρήση των drones στους σενάριους χώρους είναι κάτι το περίπλοκο, αλλά με το χρόνο νομίζω θα ρυθμιστεί. Θα αποκτήσουν δηλαδή ένα αέριο χώρο και θα ενταχθούν σε αυτόν. Δεν νομίζω όμως ότι η ένταξή τους θα καθορίσει το ρυθμό με τον οποίο εμείς εργαζόμαστε στο μέλλον. Τώρα, τι βήματα μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη. Εγώ εργάζομαι για ένα οργανισμό έρευνας και ανάπτυξη που βασίζεται σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε κατά κάποιο τρόπο ο στόχο μου είναι ανοιχτό. Ο ρυθμό τη καινοτομία προποθέτει χρηματοδότηση ευρωπαϊκή και οι δραστηριότητε οι μελλοντικέ στον τομέα τη ψηφιοποίηση τη αεροπλοεία θα είναι σημαντικό στοιχείο. Τώρα κατά πόσο μπορούμε να πάμε σε μεγάλη κλίμακα, σε μαζική κλίμακα, αυτό θα μπορούσε να γίνει, αλλά θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο βαθμό ολοκλήρωσης και συντονισμού. Και προσπαθώ αντικειμενικά να πω ότι οι εταιρικέ σχέσεις που έχουμε συνάψει ως ΣΕΖΑΡ στην Ευρώπη είναι ένα πολύ καλό μοντέλο για το πώς δημιουργούμε συνενέσεις για τις προτεραιότητες, για τις ανάγκες χρηματοδότησης και αυτή είναι η προσέγγιση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλενέρ, πολύ σύντομα. Ναι. με αντίστροφη σειρά να απαντήσω, Βυρκόνεν, για το πώς θα άρουμε τους φραγμούς και να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις. Η ψηφιακή αγορά είναι σημαντική, αλλά όταν άπτεται της πραγματικής οικονομίας, εκεί ακριβώς θα πρέπει να δουλέψετε για να απαλείψετε τους φραγμούς. Η αεροπλοεία είναι μια επιτυχής, ένας επιτυχής τομέας, ένα success story, γιατί όλοι μπορούν να πετάξουν, όλοι έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες. Και η ψηφιακή οικονομία ακολουθεί αυτομάτως και εκεί θα πρέπει να απαλείψουμε φράχμους και είναι σημαντικό όπου υπάρχει νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εφαρμόζεται και οι χώρες μέλη θα πρέπει να παρεμποδίζονται όταν αρχίζουν να ακολουθούν πρακτικές προστατευτικές. Για τον κύριο Κοκ, για το κατά πόσο χρειαζόμαστε ρυθμίσεις για τις ολοκληρωμένες μεταφορές. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποιος προσπαθεί να το αποτρέψει. Και αυτό που βλέπουμε στον σιδηροδρομό ή στις δημόσιες μεταφορές όπου έχουμε μονοπόλια, όπου έχουμε τόσο πάνω οργανισμού που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να μοιραστούν πληροφορίες ε, όσον αφορά την εκδοσή στήριων κτλ. Εκεί ακριβώς θα πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις για την διόρθωση της αγοράς. Αυτό θα ήταν η συμβουλή μου προς όποιον ενδιαφέρεται. Και για τον κύριο κάμπ αυτά που είπε, να απαντήσω για την λήψη αποφάσεων η οποία είναι αργή. Αυτό είναι το τίμημα της ειρήνης στην Ευρώπη. Νομίζω, αλλά δεν έχει τόσο να κάνει με το ρυθμό λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις οικονομικές ρυθμίσεις όπου ο ρυθμός είναι ε, επαρκής, εμένα με ανησυχεί περισσότερο, περισσότερο ο ρυθμός επιβολής και εφαρμογής. Δηλαδή, αν χρειάζονται 5-6 χρόνια για να εφαρμοστεί κάτι το οποίο αποφασίστηκε, ε, κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, για μας συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα να πω, με λύπη δυστυχώ ότι ναι, πράγματι έχουμε μια νέα εξέλιξη και είχαμε μια αναφορά στον τύπο γι' αυτό, ότι μετά από τρία χρόνια έρευνας, η Κομισιόν φαίνεται να μας λέει ότι δεν υπάρχει ε, ενδιαφέρον να διερευνήσει αυτή την υπόθεση και την απορρίπτει, κάτι το οποίο για μας είναι απαράδεκτο. Αν υπήρχε απόφαση επί της ουσίας να το δεχτώ, όμως απόφαση μετά από τρία χρόνια απορριπτική, μετά από διάφορα παράνομα, ε, παράπονα, γιατί δεν παραπονιόμαστε μόνο εμείς, αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχει και συνέχεια το θέμα και ελπίζω να έχουμε την στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κλενέρ. Μπορούμε να τους χειροκροτήσουμε τους εισηγητές μας για τις εισηγήσεις τους. Σας ευχαριστώ κύριε Κλενέρ, κύριε Μπατσελόρ και κύριε Μουσκέ. Πάμε τώρα στις τέσσερις ευρωπαϊκές νεόφυτες της startup που κέρδισαν το βραβείο για την κινητικότητα. Ελάτε εδώ να καθίσετε, νεόφυτοι και νεόφυτες, καθίστε. Μη φοβάστε, ελάτε εδώ δίπλα μου, δεν θα αγκωνώ. comment ça va depuis euh, février dernier? Τι γίνεται λοιπόν από τον περασμένο Φλεβάρι, πώς πάνε τα πράγματα, καλά, καλά, ωραία. Τρία λεπτά έχετε ο καθένα σας και η καθεμιά σας, λέει πρόεδρος, για να μας παρουσιάσετε τις νεόφυτες σας επιχειρήσεις. Ξεκινάμε την Cargo Next, ο Rolf Dieter Lafrentz. Έχετε το λόγο, κύριε Λαφρέντς, τρία λεπτά να μας παρουσιάσετε ακριβώς την νεόφυτη σας ε, επιχείρηση και μας πείτε και από πού κατάγεστε, είναι σημαντικό. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Μικροφώνο δυστυχώς ο κύριος ε, Ρολφ Τίτερ Λαφρέντς. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ιδρυτή και πρόεδρος της CarConnex από τη Γερμανία, εμείς δημιουργήσαμε το πρώτο FES ε, δίκτυο οχημάτων, μειώνοντας ακριβώς τις κενές μετακινήσεις που έχουν τεράστιες επιπτώσεις όσον αφορά τους ρήπους και τις εκπομπές τους. Η αγορά αυτών των οχημάτων, τα HGV, είναι τεράστια εμπλέκονται εδώ πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε και πολλά δισεκατομμύρια χιλιόμετρων που διανύουν αυτά τα χιλιόμετρα ετησίω. Έχουμε σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Καταρχάς το κόστος συναλλαγών και το άλλο μεγάλο πρόβλημά μας, σύμφωνα με μια ομάδα παροχής συμβουλών της Βοστόνης, είναι το ότι 25% των μετακινήσεων των ταξιδιών αυτών είναι κενά. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει στο να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, δηλαδή δημιουργώντας ένα δίκτυο εφιών μεταφορών. Θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να το κάνουμε σαν το Uber, όπου μπορείτε με ένα κλικ του ποντικού να παραγγείλετε ένα μεταφορέα, όπως κάνετε με ένα όχημα του Uber. Για το δίκτυο αυτό έχουμε δημιουργήσει αλγόριθμους που μαθαίνουν και μπορούν να κάνουν προβλέψεις ώστε να συνδυάσουν τη ζήτηση με την προσφορά ώστε να χρησιμοποιούμε ακριβώς το δυναμικό πιο αποτελεσματικά, να αποφύγουμε τα κενά ταξίδια, να μειώσουμε την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τους δρύπους. Όλα αυτά πάνε πολύ καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που κερδίσαμε αυτό το βραβείο για τις νεόφυτες. Είχαμε και άλλες ε, βραβεύσεις και είχαμε 400% αύξηση στον όγκο των μεταφορών μας. Άκουσα προηγουμένως ότι χρειαζόμαστε ένα αριθμιστικό πλαίσιο, χρειαζόμαστε ψηφιακά έγγραφα, χρειαζόμαστε εναρμονισμένη νομοθεσία στην Ένωση. Συμφωνώ και θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να έχετε κατά νου το εξής. Όταν δημιουργεί κανείς μια νεόφυτη επιχείρηση ψηφιακή, είναι σαν να, κάνει, σαν να συμμετέχει σε ένα αγώνα Φόρμουλα 1, όπου έχουμε τεράστιους ανταγωνιστές, Amazon, Alibaba, Uber, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παγκοσμίω. Χρειαζόμαστε λοιπόν ανοιχτέ αγορέ, χρειαζόμαστε χρήματα, το πρόγραμμα Horizon, ορίζοντα τη Ένωση είναι πολύ καλό και χρειαζόμαστε και παροχή εξωτερική ε, συμβουλών για να εφαρμόσουμε κάποια από αυτά τα προγράμματα. Επίσης πρέπει να μειώσουμε και τις προθεσμίες. Θα πρέπει να λύσουμε το ρυθμιστικό χειρόφρενο, γιατί καμιά φορά ε, η νομοθεσία είναι πολύ δύσκολη για μας. Ευχαριστώ. Κοκοντή από τον κύριο Βενσάν θα ακούσουμε τώρα την παρουσίαση. Από την κυρία μάλλον. Έχω συνειδρήσει εγώ το κοκολί. Είναι μια υπηρεσία που απευθύνεται στους ιδιώτες επαναφευρίσκουμε τη μεταφορά αγωθών, κυρίως των μεγάλων αγαθών για τους ιδιώτε, των μεγάλων πορευμάτων. Για τους ιδιώτε είναι πολύ ακριβό να μεταφέρουν ένα αγαθό που είναι μεγάλο και βαρύ. Α καναπέ, μια κιθάρα, λάστιχο, ένα ποδήλατο. Μπορεί να κοστίσει δεκάδε ευρώ, εκατοντάδε ευρώ και καμιά φορά δεν υπάρχει λύση ε, μεταφορά με τα παραδοσιακά μέσα. Εμεί τι κάνουμε στο κοκολί συσχετίζουμε αυτού που έχουν ανάγκη να στείλουν αντικείμενο με εκείνου που έχουν συγκεκριμένη διαδρομή που θα ακολουθήσουν και έχουν ε, θέση ε, στόχημά του. Μπορεί να γίνει μεταφορά με φορτηγάκι, με λεωφορείο, με τρένο, με γιοταχή. Δεν υπάρχει όριο όσον αφορά ε, τη διαδρομή που εκτελείται. Ποιο είναι το όφελο. Επιτρέπουμε μια φθηνότερη παράδοση, ε, εξοικονόμηση αριθμού χυμάτων στο δρόμο, διότι οι περισσότεροι πελάτε μα. Ε, δεν χρησιμοποιούν παραδοσιακά μετα, ε, αν δεν είχαν παραδοσιακά μέσα, χρησιμοποιούν το χυμά του. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την κυκλοφορία. Ε, ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν το αυτοκίνητό του καθημερινά, πάνω από 60%. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε μια απάντηση σε αυτό το θέμα. Εκεί που υπάρχουν λίγοι, κυρίως κινούνται αυτοί που μεταφέρουν ε, από 3 κιλά μέχρι 70 κιλά. Υπάρχουν παραδοσιακές λύσεις, FedEx, ε, UPS, DHL. Όταν πάμε όμως στα μεγάλα αντικείμενα, όπως τις ε, μετακομίσεις, και κάποιος θέλει να στείλει μεγάλο αντικείμενο ή να κάνει μικρή μετακόμιση, μόνο για μεγάλες μετακομίσεις υπάρχουν λύσεις, για μια μικρή τέτοια μεταφορά μεγάλου αντικειμένου είμαστε εμείς. Θέλουμε να είναι πιο εύκολη και οικονομική λύση για όλους. Ανακοίνωση, μηνύματα ανταλλάσσουμε και μέσω ασφαλούς τρόπου γίνεται η πληρωμή και υπάρχει και ασφάλιση που καλύπτει όλα τα αγαθά, όλα τα προϊόντα που μεταφέρονται αν τυχόν συμβεί κάτι. 4.000 άτομα έχουμε που συνεργάζονται. Είναι πολύ ικανοποιημένοι άνθρωποι, οι πελάτες μας. Και τι περασπιζόμαστε. Την οικονομία, την οικολογία και πραγματικά είναι καινοτόμα η λύση μας μέσω της ψηφιοποίησης των μεταφορών και του συσχετισμού των ανθρώπων. κινούμεθα στην ε, Γαλλία, είμαστε Γάλλοι, κινούμεθα στην γαλλική αγορά. Θέλουμε να προωθήσουμε την κοκολή και στην Ευρώπη, διότι δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκή κλίμακα αυτή η λύση και νομίζω ότι καλύπτει ε, τις ανάγκες των ιδιωτών και παραδείγματο χάρη μεταφορές συνοριακές μεταξύ Γαλλίας, ε, Βελγίου, Ελβετίας, Ισπανίας κλπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βανσά. Την Πολάλεν, της Mass Global. Ε, μπορείτε να μας παρουσιάσετε τη Mass Global. Έχετε το λόγο. Oh, sorry. Uh, for the to... Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να παριστάμεθα. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να θέσουμε το ερώτημα, το βασικό. Να ρωτήσουμε τους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουμε για να παρτηθείτε από τη χρήση του οχήματό σα. Δεν μπορεί να υποχρεώσουμε κανέναν να το κάνει αυτό. Πρέπει να βρούμε καλύτερε εναλλακτικέ. Πιο επιθυμητέ εναλλακτικέ. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει το μέσο κόστος είναι πάνω 500 ευρώ όσον αφορά τον ιδιοκτήτη γεωταχή αλλά οι, τα, τα που χρησιμοποιούνται κατά τον κύκλο ζωής 4% και το κόστος των μεταφορών κυρίως βαρύνει τα ιδιώτα κυρίως τα ιδιώτα χρησιμοποιούν. Με τα ιδιώτα μπορούμε να κάνουμε άλματα όσον αφορά ε, τις μεταφορές. Και έχουμε το πρόβλημα της ρήπανσης που προξενούν τα ιδιώτα Τι θέλουμε να προσφέρουμε αντί να έχουν γεωταχή στη διάθεσή τους, θέλουμε να έχουν ελεύθερη κινητικότητα. Σε όλο τον κόσμο, με διάφορα μέσα. Έχουμε το WIM. Λοιπόν, θέλουμε να συνδυάσουμε όλες τις μεταφορικές υπηρεσίες, δημόσιες μεταφορές, ταξί, αυτοκίνητα, μαζικές μεταφοράς, ε, ποδήλατα σε μια ενιαία λύση και ταιριάζουμε τις προσφορές μας, τις ανάγκες του ε, ιδιώτη ε, σε μηνιαία πακέτα. WIM μας λένε, έχουμε, είμαστε φιλανδική εταιρεία, είναι λίγα τα χρόνια από όταν έχουμε ιδρυθεί. Είμαστε στη Φιλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο. 15,4 εκατομμύρια ευρώ έχουμε δεχτεί επενδύσεις και κερδίζουμε έδαφος ε, και κερδίζουμε και βραβεία, όχι μόνο για την κινητικότητα, αλλά λόγω του σχεδιασμού των υπηρεσιών που παρέχουμε. Προσπαθούμε να έχουμε μεγαλύτερη διασυνδέσεις, καλύτερες διασυνδέσει για τον τελικό χρήστη. Πώς γίνεται αυτό. Συνεργαζόμαστε με παρόχους μεταφορικών υπηρεσιών που υπάρχουν, συναθρίζουμε όλες τις υπηρεσίες σε ένα νέο πλαίσιο ταξί, δημόσιες μεταφορές, ε, ποδήλατα, οχήματα και στο μέλλον και μεταφορές ε, μεγαλύτερης απόστασης. Δεν είμαστε μόνο πολυτροπικός φορέας, αλλά συναθρίζουμε όλα τα μεταφορικά μέσα. Μπορούμε να έχουμε μια περιαγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν ήδη υποδομές και προσφορά. όσοι χρησιμοποίησαν το WIM είδαν θετικά αποτελέσματα. Αυξήθηκαν οι δημόσιες μεταφορές, η χρήση δημόσιων μεταφορών. Αυτοί που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν λιγότερο τα ΙΟΤΑΧΗ. Πού μπορεί να γυρθεί η Ευρώπη. Θέλουμε να έχουμε οικοδομικούς λίθους στην Ευρώπη για να κινηθούμε μαζικά σε παγκόσμια κλίμακα. Θέλουμε να έχουμε apps ανοιχτά. Έχουμε πολύ καλές υποδομές. Έχουμε ε, περιαγωγή των δεδομένων. Αν θέλουμε να ηγηθούμε στην κινητικότητα, πρέπει τώρα να κινηθούμε και να δημιουργήσουμε τους, τα οικοδομικά υλικά για να δημιουργήσουμε αυτό το οικοδόμημα της κινητικότητας. Τι θα κάνουμε στο μέλλον. Θέλουμε ανοιχτό οικοσύστημα περιαγωγή, ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων μαζικών φορέων όπως είναι η WIM. Αυτό είναι το μέλλον, έτσι το βλέπουμε εμείς. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Τέλος, exit. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Φανταστείτε είστε στις Βρυξέλλες, φτάσατε στο σταθμό του τρένου και προσπαθείτε να έρθετε στο κοινοβούλιο, παίρνετε ένα ταξί. Και δεν υπάρχει κανείς στους δρόμους, έρχεστε εδώ αμέσως, αναπνέτε καθαρό αέρα, ανοίγετε και το παράθυρο. Δύσκολο να το φανταστεί αυτό κανείς τώρα να συμβαίνει, διότι για τους περισσότερους δεν είναι τόσο εύκολη η μετακίνηση στην πόλη, Υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, ρήπανση του αέρα, ο καθένα είναι μέσα στο αυτοκίνητό του μόνο του και αυτό είναι ανόητο πλευρά οικονομική και οικολογική. Ποιο είναι το όραμά μα, Να είναι εύκολε οι μετακινήσει εντό των ε, πόλεων. Πιο εύκολο για εσά, αλλά και για όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Τι είναι το Claxit, Είναι η εφαρμογή στη Γαλλία που αφορά τι μεταφορέ σε πόλει ε, για κοινή χρήση αυτοκινήτων Έχουμε 140.000 ε, και περισσότερες προσφορές την ημέρα και έχουμε συλλέξει 4 εκατομμύρια ευρώ. Ε, επί μακρόν παλεύουμε σε αυτό το τομέα. Από την αρχή του 2017 τελικά βρήκαμε το σωστό μοντέλο και βρήκαμε το μυστικό μας, το μυστική μας άλτσα του ΣΥΠΗΝ. Πρώτα απ' όλα ε, μία εφαρμογή κινητού που βασίζεται στα big data και σχετικές ε, διεργασίες που μπορούν να βρουν ποιες είναι οι ανάγκες σας και, και ποιοι ακυρώνουν δρομολόγια κλπ. Και, και από το Σεπτέμβριο 2018 θα μπορούμε να σας φέρουμε πίσω ε, μεταξύ αν αυτός που έχει αναλάβει μεταφέρει τελικά καιρό στο ταξίδι. Έχουμε και διάφορες εταιρείε πελάτες ε, και μπορούμε να δημιουργούμε δίκτυα εντό εταιριών ούτως τόσες συνάδελφοι να κάνουν διαδρομές μαζί και σωστή χρηματοδότηση ε, και χρηματοδότηση των μεταφορών. Οι δημόσιοι φορείς να χρηματοδοτούν αυτή τη μετακίνηση για να χρησιμοποιείται περισσότερο, γιατί έτσι και αυτή είναι η εφαρμογή μας που επικαιροποιείται κάθε μήνα. Έχουμε 150 πελάτες με ένα τέταρτο των, ε, του γαλλικού ΚΑΚ 40 είναι, μας χρησιμοποιούν και συνεργαζόμαστε με τοπική αυτοδιοίκηση σε πολλές πόλεις όπως το Παρίσι, στη Νίκαια στο... κλπ. Με τον Νότο, με τις πόλεις του Νότου. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για μας όσον αφορά την εναρμόνιση νομοθεσίας είναι σημαντικό. Αλλά πρέπει να συμμετάσχουν αυτοί που καινοτομούν στον κανονισμό περί καινοτομίας. Όλες οι εταιρείε θεωρούν ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα, η παρουσία μας εδώ. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω να είναι ένα πρώτο βήμα ενό δρόμου με μεγάλη, και να διανύσουμε μεγάλη απόσταση μαζί, διότι ε, έχουμε πολλά να κάνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Έχω κάποιες ερωτήσεις για σας. Η κυρία Ντεμόντε, επίσης. Έχετε το λόγο. Έχουν και οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ενδιαφέρει είναι η Κοκολής. Αυτή είναι η εταιρεία. Είναι ένα μέσο για παροχή υπηρεσία και για τη μείωση των εκπομπών. Και ερώτηση. Ποιος πραγματοποιεί τις μεταφορές. Αυτός που είναι επαγγελματίας, που έχει επαγγελματική δραστηριότητα, που έχει ήδη δραστηριότητα, είναι επαγγελματίας ή όχι. Μπορεί να είναι καλές πρακτικές αυτές, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε και διάφορες νομοθεσίες. Στην Ιταλία προβλέπεται ένα πλαίσιο όσον αφορά το πότε γίνεται κανείς επαγγελματίας και πότε περιστασιακά ασκεί κάποια δραστηριότητα. Αυτή είναι η ερώτηση πρώτη. Η δεύτερη. Είδα θετικά αποτελέσματα αφού νικήσατε και, το, και γι' αυτό νικήσατε και πήρατε το βραβείο. Τι γίνεται στον αφορά ανταγωνισμό με τα ελαφρά οχήματα μεταφορικά. Αυτοί πώς δέχτηκαν ε, αυτή την είδηση στη δημιουργία της εταιρείας σας και την όλη κατάσταση. Ευχαριστώ κυρία Ντεμούντε. Κυρία, Μέσνερ, είχε στήσει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Startups, klingt alles total spannend. Also zunächst mal ε, Πολύ ενδιαφέροντα, συναρπαστικά θα έλεγα αυτά που ακούσαμε. Ε, έγινε και αναφορά στο Αμβούργο, θα ήθελα να ξέρω περισσότερα γι' αυτό, διότι είναι η δική μου εκλογική περιφέρεια. Κάποια ερωτήματα. για τα ηλεκτρονικά ψηφιακά έγγραφα. Ε, πώς το καταφέρνετε αυτό επίσης με τα φορτηγά ε, πώς μπορείτε να αποφύγετε δηλαδή αυτά τα διάφορα βήματα για να, για να γεμίσετε τα φορτικά και από την κοκολή τώρα είναι κρίμα που το 2020 είναι η ημερομηνία αυτή ε, η προθεσμία θα ήθελα να σας χρησιμοποιήσω ήδη από του χρόνου τις υπηρεσίες σας. Ε, όλες οι εταιρείε ε, που λένε ότι πρέπει να έρθουμε καλύτερα σε επαφή απευθείας με τον πελάτη ε, διότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστευτικότητα. Πώς θα συνεργαστούν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Και την κυρία Πολάινεν Πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, πολύ καλή ιδέα. Κάνετε κάτι το οποίο ονειρεύονται οι ευρωβουλευτές εδώ και χρόνια, ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Έως τώρα μας έλεγαν ότι αυτό δεν γίνεται, διότι οι εθνικοί συντηρόδρομοι δεν το θέλουν. Συνεργάζονται οι εθνικοί συντηρόδρομοι μαζί σας, όμως εκεί όπου ε, επιχειρείτε, διότι είναι ένα πρόβλημα αυτό και στον εκπρόσωπο της Κλάξιτ. Είπατε ότι έχετε δεσμούς με τις τοπικές αρχές. Αυτό αποτελεί μέρος του UPNV. Πολλές από τις τοπικές αρχές θέλουν λιγότερα οχήματα, θέλουν περισσότερες δημόσιες μεταφορές και θα μπορούσε να μπει σε αυτή την κατηγορία. Πολύ γρήγορα παρακαλώ γιατί είναι και έχουμε και μετά συζήτηση. Κύριε Κόχ, όσο γίνεται πιο σύντομα, συγχαρητήρια σε όλους τους κατόχους, στους ε, βραβευμένους όπως επιπτώσει. Τώρα τα συστήματά σας λειτουργούν εθνικά, διασυνοριακά. Μήπως θα πρέπει για να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα να υπάρξει μια εναρμόνιση των κανόνων σε ό,τι αφορά την μισθοδοσία, τις, ε, ε αργίες, τις διακοπές λοιπά Τις άδειες Ευχαριστώ κύριε Κορ. Τώρα έχετε ένα λεπτό ο καθένας για να απαντήσετε από τη startup. Δεν είναι και άσχημα. Λοιπόν. Ναι, το ηλεκτρονικό έγγραφο για τα φορτηγά. Ακούστε, για την ώρα οι ίδιοι οι φορτηγατζίδες ε, παίρνουν φωτογραφία και τη στέλνουν μέσω mail. Οπότε δεν έχουμε ακόμα τις άδειε τις ηλεκτρονικές. Χρειαστούμε αυτά τα στοιχεία. Ε, για την ώρα το γραφείο είναι και το ήρω και θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό στο μέλλον. Τώρα προσπαθούμε να προγραμματίσουμε τα πράγματα με αλγόριθμού, διότι όταν εμεί πάμε από το α στο το β, μετά πρέπει να πάμε από το β στο γ, από το γ στο δ, δηλαδή πρέπει να έχουμε τα δεδομένα στη διάθεσή μας το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουμε να αρμονίσουμε, να οργανώσουμε όσο γίνεται καλύτερα τι μεταφορέ μα. Ό,τι φορά την αρμόνιση, ε, η κάθε χώρα ε, πραγματικά στην οποία επιχειρούμε είναι ένα μικρό θαύμα. Κάθε φορά πρέπει να βρούμε νέους ε, νομικούς, νέους δικηγόρους, και είναι δύσκολο με του μη εναρμονισμένου κανόνε. Οπότε χρειαζόμαστε την αρμόνιση. Ναι, για ένα λεπτό παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Για να απαντήσω ε, στο πρώτο ερώτημα. Αυτοί που χρησιμοποιούν την, το κοκολί για τη μεταφορά των ε, αντικειμένων είναι ιδιώτε. Ε, έχουμε, μοιραζόμαστε τα έξοδα, μοιραζόμαστε το αυτοκίνητο, δεν μπορεί κάποιο να, να αποκομίσει όφελο. Από εκεί και πέρα είναι λίγο μια φαιά ζώνη από πλευράς. Υπάρχουν προβλήματα νομοθεσίας. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νομοθεσία στη Γαλλία εντό τη οποία προσπαθούμε να κινηθούμε. Αλλά γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλουμε να επεκταθούμε στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, θα ήταν καλό να υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία κοινή για όλου. Ε, τώρα είναι θέμα μέσων ε, η διεύρυνσή μα, ε, πρέπει να μπορέσουμε να επενδύσουμε, να προσλάβουμε τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε πάντως σε νομικό επίπεδο το European το βραβείο αυτό μας μας επιτρέπει να έχουμε μια νομική ε, συνδρομή που θα μας επιτρέψει και με τη σειρά μας από εκεί και πέρα να πλαισιώσουμε καλύτερα την επέκτασή μας στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως λειτουργεί ήδη από τη Γαλλία με τις διασυνοριακές ε, χώρες. Ευχαριστώ. Η Ζωανά τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αντιμετωπίζουμε ζητήματα με όλα τα μεγάλα μονοπόλια στον τομέα των μεταφορών, εθνικοί σιδηρόδρομοι, ε, αλλά και υπηρεσίες ε, που έχουν μεγάλες συμπράξεις. Όλοι χρησιμοποιούν ε, την δεσπόζουσα θέση τους και δεν ε, ανοίγουν εύκολα την αγορά. Έχουμε όμως και καλά παραδείγματα από τη Φιλανδία. Ε, το Φιλανδικό Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνίων ε, δείχνει το δρόμο και τροποποιεί την νομοθεσία περί μεταφορών και με την νέα αυτή νομοθεσία προβλέπεται ότι όλες οι, όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών θα ανοίξουν τις πληρωμές όχι μόνο τα στοιχεία για τις μεταφορές αλλά και για τις πληρωμές προς τους τρίτους ε, παρόχους υπηρεσιών, όχι μόνο δηλαδή για μας, αλλά και για τους συναγωνιστές μας, ε, ανταγωνιστές μας μάλλον. Ε, οπότε ζητούμε, ζητούμε συμπράξεις, εταιρικές σχέσεις, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τέτοιες υπηρεσίες για τους πελάτες μας. Για ένα λεπτό παρακαλώ και εσείς. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, το carpooling θα πρέπει να αποτελεί μέρος των δημοσίων μεταφορών. Αυτή είναι, αυτό είναι το όραμά μας, έτσι το βλέπουμε εμείς. Παραδείγματο χάρη αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για, την, για τα προάστια σε, σε ζώνες που είναι μακριά από το κέντρο. Ε, στη Γαλλία έχουμε συνεργαστεί συχνά με τέτοιες ε, περιοχές ε, και ήδη έχουμε δεκαπλασιάσει τον πληθυσμό που εποφελείται από αυτή την υπηρεσία και έχουμε διαιρέσει τον, προπολογισμό δια 8. Εμείς έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή από ότι ο δημόσιος τομέας σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι σημαντικό βεβαίως να είναι τυποποιημένη, να είναι εναρμονισμένη η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην καλή αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι, γκρίζας, είναι μια γκρίζα ζώνη. Θέλουμε να υπάρξει μια ρύθμιση και για τις αρχές αλλά και για τις εταιρείε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και στους τέσσερις να τους, να χειροκροτήσουμε. Είναι τέσσερις πρώτοι νικητές και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Συνεχίστε ε, το ευρωπαϊκό σας, την ευρωπαϊκή σας τουρνέ. Και τώρα οι τρεις επόμενοι ομιλητές, ε, παρακαλώ. Ο κύριος Μάρτιν Ντόρσμαν πρώτα. Ο Ζων Λουίζε Γόμ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 Θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στον Μάρτιν Ντόρσμαν, είναι Γενικό Γραμματέα τη Ένωση ε, ε, ε, της, Επιτροπής Ευρωπαίων Πλειοκτητών να μας πείτε την άποψή σας για τις μεταφορές. Έχετε το λόγο ευθύς αμέσως. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Καλή σας μέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε κάλεσε την ΕΞΑ. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση, πέντε λεπτά ελπίζω, λέει ο κ. Ντόρσμαν, για την ψηφιοποίηση στον τομέα των μεταφορών. Θα αναφερθώ ε, στην τηλεπικοινωνία μεταξύ του πλοίου και του λιμανιού, όταν το πλοίο εισέρχεται στο λιμάνι, διότι είναι ένα, τα ζητήματα που μας προσχολούν και εδώ το Κοινοβούλιο για την εξάμιση προς, πούμε 21 ενώσεις πλειοκτητών ευρωπαϊκών χωρών και της Νορβηγίας δημιουργήθηκε το 1965, η βάση μας είναι στις Βρυξέλλες. Εάν δούμε τώρα την ψηφιοποίηση στον τομέα των μεταφορών και των πλοίων, ε, και δεν είναι μόνο τα πλοία, για τα πλοία όμως πρώτα, ποιος είναι ο σκοπός, ποιος είναι ο στόχος της ψηφιοποίησης. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι ένα μέσο για να πετύχουμε κάποια αποτελέσματα. Ένα σημαντικό στόχο λοιπόν είναι να μειωθεί το διοικητικό άχθο ε, στον κλάδο μα όταν φτάνει ή φεύγει ένα πλοίο από το λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα λιμάνι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε ε, να μειώσουμε το κόστο ε, του εξωτερικού εμπορίου τη Ένωση, αλλά και του εμπορίου εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα για τι μικρέ ε, αποστάσει τα μικρά δρομολόγια τα θαλάσσια Υπάρχει ήδη μια σημαντική βελτίωση, έχουμε μια πολύ καλή θέση στην αγορά. Θέλουμε να βελτιώσουμε αυτή τη θέση για να μειωθεί και το περιβαλλοντικό άχθος. Υπάρχει μια άλλη σημαντική πτυχή, η μείωση της ε, επιβάρυνσης ε, ε, των, του προσωπικού του πλήρου πληρώματος περνούν 2 με 3 ώρες τη μέρα με διοικητικά ζητήματα. Αυτό θα αυξήσει και την ικανοποίηση στον χώρο εργασία αλλά και την ασφάλεια. Έτσι μπορεί δηλαδή, το πλήρωμα να κάνει άλλα πράγματα που είναι σημαντικά για τα ζητήματα ασφαλείας. Τώρα, όταν μιλάμε για την ψηφιοποίηση, πρέπει να ξέρουμε ότι τα πλοία αποτελούν μέρο μια ευρύτερη αλυσίδα. Ε, η ψηφιοποίηση σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του του συνόλου τη αλυσίδα. Αυτό σημαίνει επίση ότι το κόστος του εξωτερικού εμπορίου τη Ένωση ε, θα μειωθεί και του εξωτερικού εμπορίου και θα βελτιωθεί και η περιβαλλοντική απόδοση της ε, αλυσίδα. Ε, είχαμε χιλιάδες τόνους που περίμεναν πολλές μέρες για να μπουν σε ένα λιμάνι με μεγάλες επιπτώσεις περιβαλλοντικές. Τώρα, για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους όμως, πώς θα, πώς θα γίνει αυτό, διότι ωραία ακούγονται όλα αυτά. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή δεδομένων, πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τα δεδομένα μεταξύ λιμένων, μεταξύ εθνικών αρχών. Υπάρχουν εδώ κάποιες προκλήσεις. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε τα σετ δεδομένων, τα πακέτα δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε πλέον την εμπειρία ότι δεν υπάρχει τέτοια εναρμόνιση μεταξύ κρατών μελών ακόμα και μεταξύ λιμανιών στο ίδιο κράτο μέλο Ζητούνται διαφορετικά στοιχεία. Χρειάζεται ένα εναρμοσμένο τρόπο αναφορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα αρμονίσει αυτό. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη. Έχουμε την εμπειρία ότι αυτό οδηγεί ε, σε αρνητικά αποτελέσματα. Θα πρέπει επίσης να έχουμε ανοιχτά πρότυπα, ε, τεχνολογική ουδετερότητα, ιδιαίτερα όταν επικαιροποιούμε τα συστήματα. Αυτό πρέπει να γίνεται με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να συμμετάσχει με τη δική του τεχνολογία και να χρησιμοποιήσει τον αρμοσμένο σύστημα. Η ανταλλαγή δεδομένων τώρα στην αλυσίδα ε, προϋποθέτει ότι θα υπάρχει εμπιστοσύνη αλλά υπάρχει ένα θέμα της διοκτησίας των δεδομένων, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα, ποιος έχει την άδεια να τροποποιήσει δεδομένα, όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν. Τώρα, κατά πόσο πάμε προς το σωστό δρόμο, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα αυτό. Ναι, και όχι. Και ναι και όχι. Αν δούμε την πρόταση για την αλλαγή τη οδηγία, ναι, πάμε προ αυτή την κατεύθυνση, όμω όμως χρειάζεται βελτίωση. Έχουμε κάποιε ανησυχίε. Ε, δεν μα ικανοποιούν κάποια από τι ε, προτάσει και κάποια από του στόχου. Δεν πάμε καλά δηλαδή, αν εξετάσω τι γίνεται με τα νέα συστήματα, τα εθνικά συστήματα τελωνίων που πρέπει να είναι έτοιμα στο 2020 και το νέο σύστημα ε, για τις αναφορές 2024. Πρώτα δηλαδή θα πρέπει να, συμμετά, να συνηθίσουμε στα εθνικά συστήματα και στη συνέχεια θα έρθει το ευρωπαϊκό σύστημα για τις αναφορές ε, όπου οι ίδιες απαιτήσει θα ζητηθούν βέβαια. Βεβαίως πάμε καλά σε ό,τι αφορά τις, ε, την οδηγία για τον λιμένα υποδοχής, την αρμόνιση των κανονισμών με τον IMO και την ηλεκτρονική αναφορές, αλλά δεν πάμε καλά σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές ε, φορολογικές αναφορές. Ε, ε, το τελευταίο που θέλω να πω τώρα, η ψηφιοποίηση είναι σημαντική, αλλά μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε και να εναρμονίσουμε τους κανονισμούς. Τα κράτη-μέλη πρέπει να δεχθούν ότι υπάρχει ένα ευρύτερο κέρδος όταν ε, ευθυγραμμίζουμε τα πράγματα και εναρμονίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο των διαφορών συστημάτων αναφοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντόρσμαν. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον Ζων Λουίζε ο οποίος είναι διευθυντής, γενικός διευθυντής της ΑΡΠΗΣ, ε, Δεν ξέρω αν έχουμε διακαθυστέρηση. Παρακαλώ για το λόγο. Ναι, θα παρουσιάσω πρώτα τη συνεργασία που υπάρχει ε, για τον Άνω Ρήνο. Ποιος είναι, τι είναι ο Άνω Ρήνος. Ε, πρόκειται για το κομμάτι εκείνο του Ρήνου που βρίσκεται ε, στην Πάδη Βουρτεμβέργη, Ρινανία, Αλσατία ε, και, την Ελβετία όπου εμείς εκεί έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα συνεργασίας το οποίο όπου συμμετέχουν μάλλον νέα ευρωπαϊκά λιμάνια. Αρκετά παραδειγματική, ε, είναι τριεθνής, 1.300 εταιρείε συμμετέχουν, εννέα hub ε, ε, multimodal, 50 ε, εκατομμύρια τόνοι μεταφορών, δύο επίπεδα συνεργασίας μας βοήθησαν τα, τα προγράμματα και τα SEF για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη συνεργασία. Ποια ήταν η διαπίστωση αρχική. Διαπιστώσαμε ότι σε επίπεδο τεχνολογιών επικοινωνίας υπήρχε πολύ λίγη ολοκλήρωση, πολύ λίγη κοινή προσέγγιση και αυτό οδηγούσε σε ζητήματα, σε προβλήματα ε, συμφόρησης και στα διάφορα τέρμιναλ, στους θερματικούς έπρεπε να λειτουργήσουν αυτά αποτελεσματικά. Αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις, δημιουργεί κόστος, αντιλαμβάνεστε ότι όταν σε ένα τερματικό μια ομάδα είναι έτοιμη ε, να υποδεχθεί ένα πλοίο και το πλοίο φτάνει δύο ώρες αργότερα, τα πράγματα δεν είναι καλά. Τέλος, ε, χρειάζεται αποκέντρωση της ανταλλαγής δεδομένων, ε, χρειαζόταν μεταξύ των κρατών μελών και, και των χωρών εκτός Ευρώπης όπως η, η Ελβετία που προκύπτουν και τελωνιακά ζητήματα σε σημεία όπου τρεις χώρες είναι πολύ κοντά αυτό δημιουργεί και άλλε καθυστερήσει και άλλο κόστο. Ε, εξού λοιπόν και αυτή η ιδέα αυτού του συστήματο διαχείριση τη κυκλοφορία. Βλέπετε εδώ βεβαίω ε, κάποιε οθόνε που δεν είναι και τόσο καθαρέ, Τι θέλουμε εδώ. Ε, θέλουμε κάποιο να μπορεί να κλείσει ένα σλότ σε κάποια terminals, αλλά να, να υπολογίσει το σύστημα εάν αυτά τα σλότ είναι συμβατά μεταξύ του με βάση τα container τα οποία θα πρέπει να περάσουν και με βάση τον χρόνο διαδρομής μεταξύ των διαφόρων terminals. Αυτό υπολογίζεται ε, και πρέπει να το πω αυτό μέσω ενό άλλου project που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το River Information Service πριν υπήρχαν βεβαίω τέτοια συστήματα που κλείναμε κάποια σλότ, όμω ήταν τηλεφωνικό το σύστημα αυτό. Έλεγε ο καπετάνιο, ε, βρίσκομαι στο τάδε σημείο, ε, θα φτάσω στο Στρασβούργο περίπου σε δύο ώρες και μετά βέβαια διαπιστώναμε ότι ήταν 50 χιλιόμετρα ε, πιο κάτω και το έλεγε για να κλείσει το θέση πριν από τον συνάδελφό του. Ε, λοιπόν, αυτό το σύστημα είναι επιχειρησιακό πλέον σήμερα. Ε, μας επιτρέπει χάρη στον εντοπισμό στο πραγματικό χρόνο και τον χρόνο, την εποχή του χρόνου καθυστέρηση, να ξέρουμε ποιο θα είναι ο χρόνο άφηξη και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για την επεξεργασία, για τη διαδικασία, όπω Ε, αυτό το σύστημα λειτουργεί και στα τρία σύνορα, αρχίζει να λειτουργεί και στο Στρασβούργο και θα επεκταθεί στο σύνολο των εννέα πλατφορμών. Έχουμε επίση διαπιστώσει ότι μπορεί να επεκταθεί, αν χρειαστεί, και για κυκλοφορία πιο συμβατική και για τα πετρελαϊκά τέρμιναλς αλλά και για επιβατικά πλοία και γερόπλια. Λοιπόν, ποιε είναι τώρα οι δυσκολίε, τι μάθαμε κατά τη διάρκεια αυτού του project. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να υποτιμάει κανεί ότι εδώ δημιουργούμε μια κοινότητα μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν διαφορετικέ προσδοκίε και σε πολιτισμικό επίπεδο υπάρχουν διαφορά. Άλλοι είναι δημόσιοι φορεί, άλλοι είναι ιδιωτικοί, άλλοι είναι ιδιωτικοί. Όλοι αυτοί πρέπει να συνεργαστούν. Εξού λοιπόν και μια προσέγγιση κλασική στον τομέα της πληροφορικής, ευέλικτη, που επιτρέπει να πάμε προς την επιτυχία, διότι δεν μπορούμε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το προϊόν, ε, χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται ενέργεια, ε, η πλατφόρμα πρέπει να είναι τελώς ουδέτερη, αυτό είναι κάτι το οποίο το ζήτησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ουδέτερη η πλατφόρμα αυτή, γιατί, διότι ανταλλάσσουμε δεδομένα. Κάποιος που έχει ε, όλα τα όλη την κυκλοφορία ε, στο, μπροστά στον, ε, τον ε, κοντέινερ στην, ε, στην οθόνη του, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει με αυτό. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί σε επίπεδο ασφάλεια και ιδιωτική ζωή και να υπάρχει ένα interface, μια διάδραση με άλλα συστήματα. Εκεί που υπάρχει ένα αίτημα, και εδώ συμφωνώ με τον συνάδελφο προηγουμένω, ότι υπάρχει, υπάρχει ένα αίτημα για έναν ορισμό των δεδομένων, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει ένα σωστό interface. Ε, διότι κάθε, κάθε επιχείρηση έχει το δικό τη σύστημα και εφόσον φτιάχνουμε αυτή την ψηφιακή υποδομή είναι απαραίτητο σήμερα να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Αυτά ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Λουί Ζερόμ και τώρα θα δώσω τον λόγο στον Ρομπέρτο Αμπόντιο ε, που είναι κλασικό διευθύντη του New Digital Business στην Eurostar. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε τους πελάτες μας σε αυτές τις νέες μορφές ψηφιοποίησης. Είναι σημαντικό μιλάμε για το μέλλον, αλλά στην πράξη όλες αυτές οι τάσεις ήδη είναι παρούσες. Και οι ψηφιακές τάσεις αποτελούν τον πυρήνα των εξελίξεων στις μεταφορές αυτή τη στιγμή και παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες για όλους μας για την, να εμπλέξουμε περισσότερους πελάτες μας σε αυτές τις διαδικασίες. Οι επιχειρήσεις θα είναι νομίζω σε, καλύτερες ε, θέσεις, σε καλύτερη θέση για να αποφεληθούν από την σχέση αυτή με τους πελάτες τους. Και αυτό έχει αλλάξει σε σχέση με από πριν 10 χρόνια ας πούμε γιατί έχουν νέε ευκαιρίε επιχειρήσει ώστε να είναι πιο επιτυχεί και να είναι πιο κοντά στου πελάτε του. Τώρα πάμε σε σιδηροδρομικέ επιχειρήσει. Ξέρουμε ότι οι επιχειρήσει μα είναι με χαμηλό περιθώριο κέρδου, πρέπει να είναι ανταγωνιστικέ, πρέπει να επενδύουν και θα πρέπει να βγάζουν χρήματα για κάθε επιβάτη που μεταφέρουν. Οπότε η ψηφιοποίηση είναι σημαντική. Αν δούμε τώρα τι γίνεται σε επίπεδο επιβατών στην εποπτεία όλων των επιβατικών ροών ανασταθμού. Αυτό είναι βασικό για να δούμε ακριβώ πώ θα κάνουμε την επιβίβαση πιο γρήγορη, ώστε και τελικά οι πελάτε να έχουν καλύτερη εμπειρία. Η ψηφιοποίηση λοιπόν μα βοηθάει εδώ για να κατανοήσουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πού βρίσκεται και από πού προέρχεται. Να μιλήσω και για τη διάδραση με τους πελάτες. Στόχος μας είναι να υπάρχει αξία, για τους πελάτες και για τους εταίρους μας. Και υπάρχουν δύο μεγάλοι πυλώνες εδώ. Οι πελάτες και τα δεδομένα. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή, τα δεδομένα που έχουμε για τους πελάτες με πιο ευφυή τρόπο. Σχεδιασμός. Πρέπει να ξεκινάμε από τον ε, πελάτη. Μπορεί να νομίζεις ότι έχει το καλύτερο προϊόν στον κόσμο, αλλά αν δεν ξεκινάει από τον πελάτη, δεν αξίζει. Είδαμε, ας πούμε, τι γίνεται με το Eurostar που ήταν ε, μια θετική εμπειρία. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί, κάνουμε τις δοκιμές μας, βλέπουμε τις απόψεις των επιβατών και προχωράμε. Και τα δεδομένα εδώ παίζουν μεγάλο ρόλο. Είναι δηλαδή σημαντικό να χαρτογραφήσουμε όλο τον κύκλο των πελατών μας, των, των επιβατών μας, για να ξέρουμε τι τους προσφέρουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η βιομηχανία των μεταφορών και η ταξιδιωτική βιομηχανία βασίζεται κυρίως στην έρευνα και στην αναζήτηση. Πρέπει όμως να δούμε και να προβλέψουμε τι χρειάζονται οι επιβάτες αυτές όταν θέλουν πούμε, να πάνε διακοπές. Γιατί εσείς σκέφτεστε πώς θα βρω ένα ε, διαμέρισμα στο Airbnb, πώς θα ολοκληρώσω το ταξίδι, πώς θα το οργανώσω κτλ. Οπότε οι ανάγκες των επιβατών και των ταξιδιωτών είναι κάπως πιο περίπλοκες από την απλή αναζήτηση και έρευνα. Και γι' αυτό ακριβώς αυτές οι πλατφόρμες μας πρέπει να χτίζονται γύρω από τους πελάτες. Δηλαδή να μην ε, παραβλέπουμε τις βασικές τους ανάγκες. Και εδώ ακριβώς η ψηφιοποίηση μας βοηθά να κατανοήσουμε περισσότερο το πώς συμπεριφέρεται ο πελάτης. Είχαμε πρόσφατα και μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση για τους ταξιδιώτες σε σχέση με το GDPR, όχι για να παρακολουθήσουμε τους πελάτες μας, αλλά για να τους προσφέρουμε κάτι πιο σημαντικό. Ξέρουμε ότι οι υπηρεσίε πρέπει να παρέχονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δευτερολέπτων, αλλιώς ο πελάτης θα φύγει. Και συνοψίζοντας για το τι προσπαθούμε να κάνουμε, στους δύο πυλώνες είναι καταρχάς ωφέλη για τους πελάτες και τους εταίρους μας, μακροπρόθεσμα, θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό και μια τελευταία διαφάνεια που έχουμε εδώ και το οποίο σχετίζεται με αυτά που είπαν οι προαλήσαντε για την κινητικότητα και τις μεγάλες ευκαιρίες για το μέλλον. Θα έχουμε μελλοντικά τις αντίστοιχες Google, Amazon και τα πλατφόρμες του κλάδου και θα πρέπει να έχουμε και τα θεσμικά όργανα, τα οποία θα διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο εδώ για την κινητικότητα, η οποία δεν αφορά μόνο το μέλλον, αλλά ήδη συμβαίνει τώρα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει εδώ να συνεργαστούμε, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας σοβαρέ, αποδεκτές προτάσει ποιοτικέ για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και η προέδρο. Ήταν ξεκάθαρα και διαφωτιστικά αυτά που είπατε Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε ερωτήσεις μετά από αυτές τις τρεις παρεμβάσεις. με κ. Κάμπ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω του τρει ομιλητέ για αυτά που είπαν. Δεν έχω ερώτηση, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Έχει περάσει ο χρόνος και μια καλωστικό δεν έχω ερώτηση. Όχι, δεν έχετε ερώτηση. Γι' αυτό πέρα το λόγο, ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους ομιλητές. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση για την ψηφιοποίηση. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και στο επανειδήν, ε, στο επανειδήν, στο χειροκρότημα για τους ηγητές μας. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Και συνεχίζουμε με τη συνεδρία, μα, με τη συνεδρία μας και κλεισμένων των θυρών με τους συντονιστές. Όσοι δεν έχετε να κάνετε ή δεν έχετε κάποια σχέση με αυτή τη συνεδρίαση, παρακαλώ να φύγετε.